Ξεκινάμε αγαπητοί συνάδελφοι γιατί έχουμε καθυστερήσει και πρέπει να τελειώσουμε 6 παρά 10. Θα ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Έχω κάποιες προτάσεις για αλλαγές. Θα ήθελα να σας προτείνω να μην συζητήσουμε τα σημεία 5 και 6 Να σας ζητήσω επίσης ε, η συνάντηση των συντονιστών να γίνει με την γραπτή διαδικασία, οπότε θα σας ανακοινώσω την επόμενη φορά τα αποτελέσματα. Σχετικά με το 5 για την ψηφοφορία CPR και το 6 ψηφοφορία για το περιφερειακό, να μην ψηφιστούν σήμερα για τους εξής λόγους. Εξώς αν η Κωνσταντς θέλει να παρουσιάσει την αιτιολόγηση της μη ψηφοφορίας. Ήδη πάντα έχουμε μία εκκρεμότητα, μακροοικονομική αιρεσιμότητα με την Επιτροπή και δεν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε για το σύνολο πακέτο στην δεύτερη ολομέλεια του μηνός Οκτωβρίου. Οπότε αν πάνε όλα καλά και αν πράγματι ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις, η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα μην γίνει το Νοέμβριο, οπότε δεν πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα. Να σας ενημερώσω επίσης ότι θα δούμε τι ε, μορφή θα πάρει η τελική συμφωνία, αν θα γίνει στην έκτακτη συνεδρίαση ε, της ε, Επιτροπής μας ή εάν θα ακολουθήσουμε τον κώδικα που ισχύει στην περίπτωση της συνομοθεσίας, οπότε θα περιμένουμε την Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Να σας ενημερώσω επίσης ότι ήδη είχαμε ένα τριμερή διάλογο για την μακροοικονομική ερεσιμότητα. Θα υπάρξει μια συνάντηση σήμερα το απόγευμα αργά με το Συμβούλιο. Έχουμε ένα τριμερή διάλογο δηλαδή σήμερα, έτσι ώστε να δούμε τι αντιδράσεις θα υπάρξουν στην πρόταση της διαπραγματευτικής ομάδας που έχει σαν βασικό στόχο την πλήρη συναπόφαση σχετικά με τις διακοπές. Λοιπόν, αυτοί είναι κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους δεν θα ψηφίσουμε για το ERDF. Πριν λίγες εβδομάδες φαινόταν ότι κάποιες ε, δυνητικές τροπολογίες στον κανονισμό σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία για τις μικρομεσές θα επηρεάσει και το Περιφερειακό Ταμείο. Και γι' αυτό το βάλαμε στην ημερήσια διάταξη, αλλά δεν έγινε αυτό, οπότε δεν υπάρχει κάτι για να ψηφίσουμε σε σχέση με το Περιφερειακό και όπως είπα δεν θα έχουμε και συνεδρίαση των συντονιστών σήμερα. Εφόσον συμφωνείτε λοιπόν με τις προτινόμενες αλλαγές, παρακαλώ να την κάνουμε δεκτή. Η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο και όπως σας είπα θα πρέπει να την τελειώσουμε στις 6 παρα 10 γιατί στις 6 ξεκινάμε τριμερή διάλογο για την αιρεσιμότητα. Τώρα, περνώ στις ανακοινώσεις της Προέδρου. Εγώ δεν έχω καμία ανακοίνωση να κάνω στην παρούσα φάση, οπότε περνάμε στο 3 που είναι η πρόταση έκθεσης του Γιάνν Όλμπριχτ για τους πόρους για ορισμένες χώρες από το κοινωνικό ταμείο. Στην ουσία δηλαδή ε, τροπολογία στον ισχύοντα κανονισμό. Ο Γιάνν Όλμπριχτ έχει το λόγο. Η έκθεσή μου, Πρόεδρε, άπτεται ενός θέματος που φαίνεται εύκολο από μακριά. Θα ήθελα όμως να κάνω ορισμένα σχόλια και να χρησιμοποιήσω την δυνατότητα που μας δίδει η παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσω και ερωτήσεις. Να προσπαθήσω να εξηγήσω ποιος είναι ο χαρακτήρας του κανονισμού. Πρόκειται για την ε, τροπολογία για τον λεγόμενο γενικό κανονισμό από το 2007 μέχρι το 2013, δηλαδή αλλαγή του γενικού κανονισμού, δηλαδή του 1083 κανονισμού του Συμβουλίου. Η τροπολογία αυτή τον κανονισμό αλλάζει τα όρια ε, για το ε, ταμείο και αυτό συνδέεται με τον έβδομο 7ος έβδομος διορθωτικος νέα στοιχεία οικονομικά. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι ανακατεύονται διαφορετικοί τρόποι χρηματοδότησης, κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί εύκολα, ίσως να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως η προέλευση αυτού του τμήματος του διορθωτικού 7 προέρχεται από τη Συμφωνία για τις Προοπτικές του Συμβουλίου και προέρχεται κυρίως για τη συμφωνία που αφορά την Βρετανική επιστροφή. Υπήρξε λοιπόν μια συμφωνία για τα νέα επίπεδα της Βρετανικής επιστροφής και μετά από όλες τις πιθανές πράξεις και υπολογισμούς ε, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει ισότητα στην αντιμετώπιση των κρατών μελών σχετικά με το τμήμα των πληρωμών ε, που προορίζεται στην Βρετανική επιστροφή. Μετά από όλους λοιπόν τους υπολογισμούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρήκε ότι υπάρχουν τρεις χώρες για τις οποίες φαίνεται ότι η ανισότητα και κατά κάποιο τρόπο η αδικία είναι υψηλού επίπεδου και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι δύσκολο βέβαια να βρεθεί μια λύση ή ήταν δύσκολο να βρεθεί μια λύση και η λύση έρχεται μέσω του EDSF. Δηλαδή η απόφαση λέγει ότι θα υπάρξει τρόπος μείωσης αυτού του ύψους πληρωμών του άδικου μέσω του κοινωνικού ταμείου. Συνεπώς λοιπόν εμείς έχουμε να κάνουμε με μία τροπολογία 157 εκατομμυρίων, 100 προέρχονται από τη Γαλλία, 20 για την Ισπανία και 30 για την Ιταλία. Όταν δείτε τις αλλαγές στον κανονισμό θα δείτε ότι οι αριθμοί διαφέρουν. Και γιατί διαφέρουν? Γιατί παραπέμπουν αυτή τη στιγμή στις λεγόμενες στις τιμές μονάδας, στις ισχύουσες τώρα τιμές μονάδας. Εγώ ε, λέγω στην έκθεσή μου, στην πρόταση, ότι στην ουσία υιοθετούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή λαμβάνουμε υπόψη τις πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την μείωση των διαφορών και των αδικιών. Ξέρετε ότι η Βρετανική επιστροφή συνδέεται άμεσα με την ΚΑΠ και αυτό έχει σημασία πολιτικά για μας. Χρησιμοποιεί το Κοινωνικό Ταμείο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καλύψει τις συνέπειες και τα συμπτώματα της Βρετανικής επιστροφής. Παρ' όλα αυτά, παρόλο το περίπλοκο του πράγματος, φαίνεται ότι είναι ικανοποιημένα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής ας συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε στη μείωση αυτής της αδικίας αν θέλετε και ελπίζουμε ότι η κίνηση αυτή από πλευράς του Κοινοβουλίου να εκτιμηθεί δε από το Συμβούλιο και από τους συναδέλφους που δίνουν μάχες για το κοινωνικό ταμείο. Δεν θέλουμε εμείς ε, να έχουμε μπλοκάρισμα από πλευράς αυτών που στηρίζουν το ε, κοινωνικό. Λοιπόν, ε, έχουμε να κάνουμε με τον 7ο διορθωτικό, μιλάμε με, για 150 εκατομμύρια και μιλάμε για τον κανονισμό 0713. Έχω εδώ την πρόταση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροπολογεί τον ισχύοντα κανονισμό. Εδώ έχω κάτι το οποίο να μου επιτρέψετε να ρωτήσω την Επιτροπή να το εξηγήσει κάπως. Δεν θα ήθελα εγώ να είμαι ο εισηγητή ο οποίος επαναλαμβάνει τις φράσεις της Επιτροπής και λέει ναι όλα ωραία. Διαβάζοντας την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε κάποιες εξηγήσεις εδώ για τις πληρωμές σε αιτήσια βάση προς το κοινωνικό ταμείο και λέγουμε εδώ ότι οι πληρωμές θα είναι 2 συν 3. Ε, Δεν έχουμε λοιπόν για το 2013, έχουμε μόνο ε, συν 3, έχουμε συν 2 για το 2013. Και ξέρουμε ότι το 12 πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και ειδικέ καταστάσεις που έχουν σχέση με Ρουμανία κτλ. Ίσως εδώ το θέμα να εκφράζει κάτι το τεχνικό το οποίο μου διαφεύγει ή να υπάρχει μια δυνατότητα μεταφοράς στο μέλλον. Αλλά ο κανόνας 1 συν 3 στον τομέα των πληρωμών δημιουργεί συγχύσεις. Δεν καταλαβαίνω. Τι, τι, τι, περί τίνος πρόκειται. Κάτι πρέπει να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ δεν πρόκειται για ανεπίσημο έγγραφο, πρόκειται για ένα έγγραφο επίσημο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο θα πρέπει να γίνει δεκτό από το Κοινοβούλιο και έχει μεγάλη σημασία σαν εισηγητής και σαν Επιτροπή να το κατανοήσουμε. Σχετικά με τους σκιώδεις έχω κάποιες πληροφορίες από τους πρασίνους και από τους σοσιαλιστές. Η Κώσταντ Σκρέλ έχει το λόγο. Ναι, ήθελα να σας πω πως ε, ο σκιώδης ηγητής μας ε, βρίσκεται στο τρένο ακόμα. Ή η συγκήτρια, η πα... ο Πατρίς Τυρολιέν. Αλλά ζήτησε να κάνω κάποιες ε, σύντομες παρατηρήσεις. Η ομάδα μας ε, στηρίζει πλήρως την έκθεση. Ε, είναι σύντομη οπωσδήποτε είναι σαφές και δεν θα καταθέσουμε τροπολογίες και νομίζω πως μπορούμε να πάμε και με αυτή την ιδέα στο σημερινό τριμερή διάλογο πως μπορούμε να πάμε στην απόφαση στην ε, συναπόφαση με μια γρήγορη διαδικασία για να μην κινδυνεύσει η πολιτική συνοχή. Νομίζω είναι μια καλή δυνατότητα για να δείξουμε στα κράτη-μέλη πώς μπορούμε να εργαστούμε με τρόπο έξυπνο και αποτελεσματικό. Στηρίζουμε λοιπόν την έκθεσή σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να υπονομεύσω την αισιοδοξία σας. Η Επιτροπή Απασχόλησης έχει ζητήσει και λάβει τη διαδικασία του άρθρου 50 για τρία άρθρα και άλλα τρία εκτιμώντας. Ελπίζω πως δεν θα υποβάλλουν λοιπόν κάποιες ε, ε, τροπολογίες. Μάλιστα, καλώς. Το, το αποσύρω, άρα μόνο η Επιτροπή μας ε, είναι, ε, έχει τη δυνατότητα να εργαστεί αποτελεσματικά. Ε, το έχουμε αποδείξει, λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, Ελίζαμπεθ, μια σύντομη παρατήρηση. Δεν είναι σαφές το τι θα κάνουμε σε σχέση με την προθεσμία για τις τροπολογίες, γιατί υπάρχει και το ζήτημα του ότι αναφέρονται συγκεκριμένες χώρες ενώ άλλες χώρες που είναι σε συγκρίσιμη κατάσταση ενώ άλλες χώρες όπως Πορτογαλία δεν αναφέρονται που θα έπρεπε να αναφερθούν γι' αυτό το συζητάμε στην ομάδα θα δούμε τι θα κάνουμε γιατί φαίνεται πως υπάρχει κάποια αυθαιρεσία στην επιλογή κάποιων χωρών και δεν είναι σαφές το γιατί έχει συμβεί κάτι τέτοιο και ίσως η Κομισιόν μπορεί να μας διαφωτίσει εδώ πέρα και να μας πείσει ε, για το ότι η πρότασή της είναι η σωστή. Εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες. Όπως ε, ήρθε δεν ξέρω αν είναι η σωστή προσέγγιση. Όπως είπαμε έχουμε μια επιφύλαξη ακόμα. Θα δούμε τώρα το εάν θα θέσουμε τροπολογίες. Επίσης έχει, υπάρχει στην ομάδα μας ε, όπως είπα μεγάλη επιφυλακτικότητα για το εάν και κατά πόσον είναι αιτιολογημένη η επιλογή των χωρών. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για την Κομισιόν να μας πείσει, αλλιώς θα καταθέσουμε τις τροπολογίες μας για τους Ευρωπαίους ε, συντηρητικούς ε, κύριος ε, Βλάσακ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω πως είμαστε επιφυλακτικοί και εμείς και σε σχέση με την έκθεση που είχα εγώ παρουσιάσει παλαιότερα που ήθελα να χρησιμοποιήσω ένα μέσο δοκιμασμένο που είχε τη χρήση και δεν θα είχε και κάποια επίπτωση στον ε, προϋπολογισμό. Αυτή ήταν η πρώτη αλλαγή του 1083 του 2006 και τώρα υπάρχει ένα νέο μέσο το οποίο δυστυχώς θα ζητάει από τα κράτη-μέλη περαιτέρω συνεισφορές. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι πως η Γερμανία θα συνεισφέρει 30 εκατομμύρια, η Γαλλία 24, η Πολωνία 4,5 για να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός. Και έχω και άλλα στη λίστα μου, οπότε θα ήθελα να ακούσω κάποια επιχειρήματα για να με πείσουν για αυτή την πρακτική. Σας ευχαριστώ, Γιώχιμ Τσελέρ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα στην ε, διαδικασία αυτή, γιατί δεν μπορώ να δω εδώ πέρα μια κανονική διαδικασία. Από ό,τι φαίνεται, μέσω μιας απόφασης κορυφής ε, υπήρξε μια παρέμβαση σε ένα σύστημα. Επιλέχθηκαν κάποιες χώρες οι οποίες ξαφνικά θα λάβουν χρήματα. Εντάξει, καταπολέμηση της ανεργίας των νέων ωραίο ακούγεται πάντα, αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω από το να δίνουμε χρήματα. Χρειάζονται και δομές και δεν το βλέπω αυτό να συμβαίνει. Ε, γιατί γενικώ ε, το θέμα είναι να δίνουμε λεφτά. Είτε μιλάμε για πρόσφυγες στην Ιταλία, είτε για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα. Λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν. Γιατί αντιλαμβάνομαι πως οι τρέχουσες υποχρεώσεις των ε, κρατών μελών Ε, υπερβαίνουν ε, κατά πολύ την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθεί. Πού θα βρεθούν τα λεφτά και αν μιλάμε και για τον κανόνα νη συν 2, από ό,τι φαίνεται τα χρήματα του 2013 αναβάλλονται για την επόμενη προγραμματική περίοδο όπου εκ των προτέρων ξέρουμε πως ε, μεταξύ ε, πραγματικών πληρωμών και υποχρεώσεων υπάρχει ήδη ε, μια ψαλίδα. Θα υπάρξει και άλλη αναβολή ή αυτά τα 150 εκατομμύρια θα βρεθούν μέσω περικοπών αλλού. Πώς θα ε, λειτουργήσει η όλη διαδικασία. Εγώ δεν, δεν έχω αντιληφθεί. Όλα αυτά βρίσκονται πίσω από ένα πέπλο. Σας ευχαριστώ που δώσω το λόγο στην ε, Κομισιόν. Ο Γιάν ε, θέλει το λόγο. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, πριν δώσετε τον λόγο στην Κομισιόν, πριν απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η... Μιλάμε για έναν διορθωτικό προϋπολογισμό, οπότε έχουμε νέα λεφτά που θα προέλθουν από τα κράτη-μέλη συγκεκριμένα ποσά από κάθε κράτος μέλος. Οπότε πρώτα απ' όλα θα ενισχύσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε αυτές τις τρεις χώρες. Δεν είναι νέες δομές. Γι' αυτό στην δική μου την έκθεση αλλάζουμε τα όρια για τα τρία αυτά κράτη-μέλη στο γενικό κανονισμό το ερώτημα της Ελίζαμπεθ γιατί αυτές οι τρεις χώρες. Η απάντηση είναι σαφής. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε και την εξήγηση της Κομισιόν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ανάλυσης ε, της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό το οποίο προκύπτει δηλαδή είναι πως η ανισορροπία μεταξύ των ε, κρατών μελών ε, βρίσκεται σε αυτά τα τρία κράτη-μέλη ακριβώς δεν είναι ότι είπαμε τρεις χώρες και όχι τέσσερις, ε, είναι οι συγκεκριμένε χώρες. Ε, όπως και η Ρουμανία και Σλοβακία με το ε, λεγόμενο ε, αντίστροφο δίκτυο ασφαλείας. Αυτή τη φορά είναι μια απόφαση του Συμβουλίου και γίνεται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Βεβαίω το σύστημα είναι αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για άλλα κράτη-μέλη. Απλά για, για να το εξηγήσω και στον κύριο Τσέλερ, αν είναι παλιά ή νέα τα Είναι νέα κονδύλια. Τα οποία θα πάνε στο... στον διορθωτικό προπολογισμό. Και έχουμε πληροφορίες πως η Κορεπέρ συμφώνησε ε, επί του διορθωτικού προπολογισμού. Οπότε μπορούμε να πάμε έτσι στον τριμερή διάλογο. Αλλά θέλω να ακούσω τι θα πει και η Κομισιόν. Δεν έχει κάποιος άλλος να πει κάτι, οπότε θα ήθελα να απαντήσει και η Κομισιόν. Όπως βλέπετε, η μοίρα αυτού του κανονισμού βρίσκεται στα χέρια σας. Πρέπει να μας πείσετε για το ότι ε, αυτές οι χώρες πρέπει να ενισχυθούν με αυτή τη διαδικασία. Και αντιλαμβάνομαι πως πρέπει να ψηφίσει μέχρι το Δεκέμβριο το Κοινοβούλιο, αλλιώς δεν έχει νόημα. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την επιπλέον ερώτηση που μου θέσατε και τα σχόλια τα οποία κάνατε. Ίσως ε, Πρέπει να ξεκινήσω ε, ευχαριστώντας την Επιτροπή σας που κινήθηκε ε, τόσο ε, γρήγορα. Όπως είπε και η Πρόεδρος προηγουμένως, ολοκληρώνεται η περίοδος η προγραμματική και επομένως φέτος στα τέλη του χρόνου θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει εγκριθεί ο κανονισμός, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και όπως είπε και ο κύριος Άλμπρεθ προηγουμένως και η Κορεπέρ έχει ήδη συμφωνήσει ε, με αυτήν την πρώτη ανάγνωση της πρότασης. Θα προσπαθήσω να προσθέσω κάποιες διευκρινήσεις, αλλά νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά σαφής κατά την άποψή μου παρουσίαση του κ. Άλμπρεχτς. Η πρόταση όντως ξεκινάει από τις συζητήσεις που έγιναν με, την, με τις χώρες ε, ε, στο Συμβούλιο του καλοκαιριού ε, και ακριβώς είχε στόχο την ε, ε, διόρθωση της κατάστασης η οποία προκύπτει και της έλλειψης ισορροπίας που προκύπτει από τις βρετανικές επιστροφές. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί μια χρηματοδοτική εξισορρόπηση βάσει και των συζητήσεων και των συμφωνιών για τις πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε ορισμένες χώρες. Οι χώρες, χώρες αυτές δηλαδή οι οποίες, ε, ε, οι οποίες ε, το θέμα έχοντας πρόβλημα μετά από τις συνολικές συμφωνίες του Ιουνίου. Η Κομισιόν θεώρησε ότι μπορούσε να λύσει, να εξισορροπήσει την κατάσταση βάζοντας επιπλέον κονδύλια ε, στην ε, καταπολέμηση της νεανικής ε, ανεργίας, θεωρώντας ότι αυτή είναι μια μεγάλη προτεραιότητα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης παράλληλα να γίνουν ε, κινήσεις ε, έτσι ώστε να είναι εμπροστοβαρής η χρηματοδότηση τέτοιων ε, προγραμμάτων και θεωρήθηκε ότι επιπλέον κονδύλια θα μπορούσαν να διευκολύνουν την καταπολέμηση της ελληνικής ανεργίας. Ιδίως εάν εάν προσθέσουμε ε, στις χώρες οι οποίες ξεκίνησαν ε, ε, το θέμα, εάν δούμε πόσο είναι αναλογικά το βάρος στις χώρες αυτές από τις βρετανικές επιστροφές. Δεν θέλαμε να αλλάξουμε υπερβολικά τον προϋπολογισμό έτσι όπως είχε τελικά συμφωνηθεί. Γι' αυτό λοιπόν καταλήξαμε καταλήξαμε σε αυτή την πρόταση για την περίοδο 7-13. Η προτινόμενη χρηματοδότηση, όπως είπα και προηγουμένως, συνδέεται με τον αντίκτυπο που έχουν στις συγκεκριμένες χώρες μέλη οι βρετανικές επιστροφές και συνδέεται επίσης και με την χρηματοδότηση που θα μπορέσουν ε, να αντλήσουν τα κράτη-μέλη από την ε, πρωτοβουλία των, ε, για την απασχόληση των νέων. Μιλάμε για τρεις συγκεκριμένες χώρες οι οποίες περισσότερο υφίστανται τον αντίκτυπο ε, των επιστροφών. Είναι αυτές οι τρεις χώρες οι οποίες αναφέρονται στην πρόταση που έχετε μπροστά σας σήμερα να απαντήσω σε ένα-δυο σχόλια όσον αφορά τις δομές που είναι ελλειπείς για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας. Νομίζω ότι ο κύριος Άλμπρεχτ ήταν πολύ ε, σαφής σε αυτό. Θα ε, πρόκειται για νέα χρήματα ε, τα οποία θα μπουν στα ήδη υπάρχοντα κονδύλια που προκύπτουν από το κοινωνικό ταμείο. Όταν και εφόσον προχωρήσει η πρόταση, η Κομισιόν θα καθίσει στο τραπέζι με τις κράτες με τα κράτη-μέλη ε, για να δουν προς τα πού θα ε, ε, στοχευθούν αυτά τα κονδύλια. Όσον αφορά το συγκεκριμένο ερώτημα για το 1 3 Ενδεχομένως δεν είναι πολύ σαφές αυτό το τμήμα του εγγράφου και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. λοιπόν, κοιτάζοντας ε, την ε, πρόταση βλέπετε τις ε, δαπάνες από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή όταν η Κομισιόν συνδέει τις πληρωμές με τα προγράμματα, δαπάνες δηλαδή επιτόπου αυτά τα έξτρα 150 εκατομμύρια για τα τρία κράτη θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ε, δαπανηθεί σε προγράμματα μέχρι το πέρας του 2015. Όμως, μετά το τέλος του 2015, οι χώρες έχουν ακόμα 15 μήνες ε, για να υποβάλουν όλα τα τελικά έγγραφα και τότε, αφού θα έχουν υποβληθεί λοιπόν και τα τελικά έγγραφα κλεισίματος των φακέλων, τότε ε, θα ε, μπορέσουν να γίνουν οι τελικές πληρωμές, δηλαδή ενδεχομένω τέλη του 2017 έως και αρχή και του 2018. Επομένως, εδώ δεν έχουμε κατάσταση 1 συν 3 όσον αφορά τις δαπάνες επιτόπου. Ε, μιλάμε για 1 συν 3 για δαπάνες από, την, ε, από το προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τα κράτη. Ε, ελπίζω ότι το αποσαφηνίσαμε, αλλά μπορώ να ξαναδοκιμάσω να σας αποσαφηνίσω ακόμα περισσότερο. Γιάννα. Θα προσπαθήσω να είμαι πολιτικός ορθός. Η εξήγησή σας για το 1 συν 3, πώς να σας το πω έτσι πολύ ευγενικά, είναι ανοιχτή. Αλλά εγώ θα ήθελα να προτείνουμε να μην το κάνουμε, να μην γίνει αυτό. Γιατί τότε οι πραγματικές πληρωμές θα γίνουν δεν θα γίνουν την επόμενη ε, χρονιά. Ε, ε, είναι σαν να έχουμε μια προγραμματική περίοδο 14-20 με 1-3, 1-4 που μπερδεύει πάρα πολύ τα πράγματα. Όλοι μας ξέρουμε ότι η μόνη δυνατότητα για το, F, για το 2007 μέχρι 2013 είναι το 1 2 Τελεία και παύλα. Δεν μπορεί να υπάρχει ένσυν 3. Αυτό που λέτε εσείς ε, είναι οι πραγματικές πληρωμές που θα γίνουν μετά το 2015. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας προτείνω, να σας συστήσω να μην βάλετε εδώ τον 1 συντρια, 3. Γιατί θα μπερδευτεί λίγο το σύστημα. Όταν ε, ε, και όταν ξεκινήσουμε πραγματικά να το εφαρμόζουμε τότε ε, θα χάσουμε τον μπούσουλα. Τον έχουμε χαμένο ήδη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ε, λοιπόν, ένα συν τρία τουλάχιστον, λέει η Πρόεδρος, να μην χρησιμοποιηθεί, τουλάχιστον με διαφορετικό τρόπο από, από αυτόν που ξέρουμε συνήθως. Ελίζαμπεθ, είναι δύσκολο το έγγραφο. Και το ιστορικό του είναι βεβαρημένο ξέρω ότι μας λείπουν χρήματα. Μα λείπουν, μας λείπουν χρήματα από τα κράτη-μέλη ε, για το τελευταίο προϋπολογισμό για το έτος 2013. Και φαίνεται ότι αυτό το χάσμα θα υπάρξει και για το 2014. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα τα οποία αναφέρονται εδώ δεν είναι διαθέσιμα γιατί δεν τα έχουν δώσει ακόμα τα κράτη-μέλη και δεν έχουν αυξήσει το αυξημένο ποσοστό το οποίο θα πρέπει να ε, καταβάλουν στον ε, ε, προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συμβαίνει για αυτό που είπα ή γιατί μεταφέρεται η πληρωμή για το 2013. Ε, δεύτερον, για πρώτη φορά... From the UK rebate and not the youth unemployment. Ε, ε, πρώτη φορά τα πρόσθετα χρήματα αφορούν την ανεργία των νέων. Ε, τώρα, ε, εάν προκύψουν αυτά τα επιπλέον χρήματα, βεβαίως, ε, αλλά τότε και η Πορτογαλία θα πρέπει να ενταχθεί στις χώρες αυτές, γιατί αν δει κανεί προσεκτικά τα αριθμητικά στοιχεία, θα διαπιστώσει ότι αντιμετωπίζει και η Πορτογαλία την ίδια κατάσταση. Και επομένως χρειάζονται χρήματα για αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό ακριβώς είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στον κόσμο την κατάσταση. Ε, γιατί δεν υπάρχει ταύτιση των στοιχείων, δηλαδή ποια ε, τα στοιχεία της δυναμικής ανεργίας ε, και τα κονδύλια τα οποία δίνονται στις συγκεκριμένες χώρες. Αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε. Επίσης, αυτό το ζήτημα της για την Πορτογαλία δεν το απήντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω πώς μπορεί. Ε, πρόεδρος, θα πάρεις το λόγο αν έχεις κάτι καινούργιο να μας πεις, Γιάννη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Επιτρέψτε μου. Πρέπει να εξηγήσουμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να συμφωνήσουν να πληρώσουν μόνο για τρεις χώρες. Δηλαδή 28 χώρες θα συμφωνήσουν ότι πρέπει να πληρώσουν για τις τρεις χώρες. Ξεκινώντας με κριτήρια νεανικής... Ε, αν ξεκινήσουμε όμως από το κριτήριο της νεανικής ενεργείας βεβαίως ε, θα προκύψουν διαφορετικά στοιχεία. Αλλά εδώ θέλουμε μόνο τις τρεις αυτές χώρες και πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι χώρες. Πρόεδρος, ναι, ε, άρα θα πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την νεανική ανεργία σε όλες τις χώρες οπουδήποτε αυτή είναι ε, έντονη και με αυτό, αλλά θα θέλουμε να μιλήσουμε για αυτές τις τρεις συγκεκριμένε ε, χώρες, οι οποίες θα πάρουν επιπλέον χρήματα που όμως θα τα δαπανίσουν αποκλειστικά για την νεανική ανεργία. Αυτά. Να σας πω ότι είναι πολύ στενό το, ε, το περιθώριο προθεσμία ε, για την, ε, για την υποβολή των τροπολογιών. Είναι ε, λίγη το απόγευμα της 17ης, είναι μεθαύριο αν θυμάμαι καλά, θα το ξαναδούμε. Το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια, το Νοέμβριο στην Επιτροπή μας. Ωραία, έληξε λοιπόν το ζήτημα αυτό και επομένως περνάμε στο επόμενο, είναι το σημείο 4, ε, έκθεση του Χέρμαν Βίνκλερ για την ευφυή εξειδίκευση. Χέρμαν, έχεις το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από το καλοκαίρι ανέπτυξα τις σκέψεις μου για την έξυπνη εξειδίκευση και τις ορισμένα ερευνητικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ενεπλάγησαν και τους εκπροσώπους Κομισιόν που βοήθησαν πάρα πολύ για το πώς θα γίνει η εφαρμογή στις ε, περιφέρειες. Νομίζω πως δεν υπάρχει πλέον εναλλακτική στην κινητοποίηση της καινοτομία στις περιφέρειες για να ενισχυθεί η οικονομική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον και νομίζω πως ε, η έξυπνη εξειδίκευση είναι ο κατάλληλος τρόπος ε, έτσι ώστε οι περιφέρειές μας να έχουν ε, οικονομική δύναμη στο μέλλον και να μπορούν να αντισταθούν και να είναι πιο ανταγωνιστικές. Βεβαίως Προφανώς υπάρχουν διάφορα εμπόδια στην εφαρμογή αυτής της ε, στρατηγικής, γι' αυτό ε, είχα, έχω συντάξει την έκθεση αυτή με τρόπο ευρύτατο και προχώρησα και πολύ πέρα από τον τίτλο και προσπάθησα να είναι και ανοιχτή για τις δικές σας παρατηρήσεις και εμπειρίες αγαπητοί συνάδελφοι έχετε όλοι πάρα πολλές και πολύτιμες εμπειρίες και οπωσδήποτε θα τις ε, καταθέσετε. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ολοκληρώσουμε την έκθεση έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε κάποιες ε, κατευθυντήριες γραμμές. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρουσίαση και έτσι θα αποκτήσετε και μια γενική εικόνα για το τι θα ήθελα να καταθέσω ως ε, τροπολογίες. Πράγματα δηλαδή τα οποία για λόγους ε, χώρου δεν χώρισαν στην αρχική έκθεση. Βλέπετε ήδη τα βασικά σημεία, δηλαδή ορισμός των σωστών προτεραιοτήτων μέσω μιας καλύτερης δικτύωσης στο επίπεδο των περιφερειών, συνέργεια μεταξύ των διαφόρων ε, προγραμμάτων δράσης και βεβαίω ε, και η εξωτερική διάσταση όπου στα σημεία 18 ε, και 19 θεωρώ πως υπάρχει ένα κενό στο κείμενο όσον αφορά την εξωτερική διάσταση. Η εφαρμογή βεβαίως δεν είναι λεπτομέρεια. Αυτό το οποίο αναμένουμε από τις περιφέρειες ε, έχει επιπτώσεις ε, και στην περιφερειακή πολιτική αλλά και διαστάσεις για την έρευνα και τη βιομηχανική πολιτική και είναι οπωσδήποτε μια μακροπρόθεσμη διαδικασία και οπωσδήποτε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και ε, λάθη. Πρέπει λοιπόν να δούμε και την εξωτερική διάσταση αλλά θα ήθελα να πω κάποια πράγματα παραπάνω γι' αυτό όμως. όλες οι περιφερειές ανεξαρτήτως του πόσο ανεπτυγμένες είναι και πόσα λεφτά περιμένουν πρέπει αυτοί, αυτούς τους όρους εξ άντε να τους δουν ως μια ευκαιρία. Δεν είναι εύκολο να βρεθούν οι προτεραιότητες. Δηλαδή πώς βρίσκει μια περιφέρεια τα συγκριτικά της ε, πλεονεκτήματα χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει πως θα φτάσει σε ένα βαθμό υπερεξειδίκευσης θα είναι αντιπαραγωγικός και βεβαίως χωρίς να ξεχνά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η έκθεση λοιπόν λέει κάποια πράγματα και γι' αυτό και πολλές περιφέρειες έχει κάποιο νόημα να πάνε προς μια κατεύθυνση υψηλής τεχνολογίας υπηρεσιών και όλο αυτού του πλέγματος όπου θα έχουμε τη λεγόμενη διάχυση της γνώσης σε περιφερειακό επίπεδο και να στοχεύσουν σε νέες αγορές. Επίσης, αξιόλογο θεωρώ πως το θέμα της καινοτομίας δεν αφορά μόνο την υψηλή τεχνολογία, αλλά αφορά παραδείγματο χάρη τον τομέα της υγείας, της δημογραφίας και τα λοιπά. Οπότε ιδεοδός θα δημιουργηθεί μια αλυσίδα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας από τη βασική έρευνα στην εφαρμοσμένη έρευνα μέχρι την ε, μεταφορά τεχνολογίας σε συγκεκριμένα πια εμπορικά προϊόντα και ίδρυση εταιριών. Θεωρώ όμως πως βασικό σημείο μιας επιτυχημένης στρατηγικής είναι έρευνα, εκπαίδευση και η διοίκηση που πρέπει να ανταποκριθεί. Πρέπει λοιπόν όλες οι περιφερειακές αρχές και φορείς να συνεργαστούν και οι επιχειρήσεις εδώ πέρα παίζουν σημαντικό ρόλο, τη δυναμική των επιχειρήσεων ε, είναι πάρα πολύ σημαντική, ότι δεν μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις, δεν θα λειτουργήσει ακριβώς γιατί εδώ πέρα πρέπει να δούμε αυτή την ε, διαδικασία ανακάλυψης και έρευνας που υπάρχει στις ε, επιχειρήσεις και βέβαια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εδώ πέρα παίζουν ιδιαίτερο ρόλο. Επίσης χρειάζεται μια νέα νοοτροπία των αρχών που πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως. Αν πάμε σε λάθος κατεύθυνση βεβαίως θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την κατεύθυνση οι περιφέρειες, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα καλό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης, δείκτες και πάρα πολλά δεδομένα, τα οποία θα είναι ιδεοδός και συγκρίσιμα μεταξύ των περιφερειών. Ένα τέτοιο όραμα βεβαίως θα υλοποιηθεί πιο εύκολα όσο είναι δικτυωμένες μεταξύ τους οι περιφέρειες μέσω παραδείγματος χάρη του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή του δικτύου ε, των επιχειρήσεων της Ευρώπης ε, ή των ε, εκολαπτηρίων των επιχειρήσεων. Επίσης σημαντικό κομμάτι είναι η εξωτερική διάσταση. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο εντός αλλά και παραπέρα και σβήνει το μικρόφωνο του μιλτή. να δούμε πώς μπορεί να συμπληρωθεί, όπως είπα, αυτή η αλυσίδα δημιουργίας αξίας. Σημαντική προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτής της ιδέας είναι η πάρα πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των φορέων των, της περιφέρειας και βέβαια αν κάποιος οργανωθεί ε, στο εσωτερικό μπορεί να συνεργαστεί μετά με άλλες περιφέρειες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα όπως το Silicon Europe αλλά κατά βάση μιλάμε για περιφέρειες που ήδη ε, είχαν την δυνατότητα συνεργασίας μέσω των λεγόμενων περιφερειών γνώσης. Αλλά πάρα πολλές περιφέρειες ε, διστάζουν να συνεργαστούν με άλλες, δεν ξέρω, ίσως ε, δεν θέλουν να ευνοήσουν τον ανταγωνισμό. Άλλες φορές δεν έχουν τη διοικητική ικανότητα. Ανεξαρτήτως τώρα του νομικού πλαισίου θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι περιφέρειες προς μια τέτοια συνεργασία και ένα 15% θα έλεγα των κονδυλίων πρέπει να κατευθυνθεί εκτός συγκεκριμένων προγραμμάτων. Θα δούμε βεβαίως αν λόγος θα γίνει στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Άλλα σημεία αναφέρθηκαν όπως εντονότερη παρακολούθηση και βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλύτερη δικτύωση, ενίσχυση της συνέργειας, εφαρμογή του ορίζοντα 2020 σε όλα τα επίπεδα. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα για τις παρατηρήσεις σας που αναμένω να ακούσω και αναμένω βέβαια και τη συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. Ο Γιάννης δεν είναι εδώ. Ο Είσαι σκιώδης πλέον, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα νομίζω για τις περιφέρειες, ειδικά σε χώρες που υπάρχει μεγάλη κρίση και η καινοτομία και η έρευνα είναι εργαλείο για να βγουν από την κρίση, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές. Ήθελα περισσότερο να εντοπίσω μερικά στοιχεία τα οποία δυσκολεύουν τις περιφέρειες ακριβώς εκείνες που χρειάζονται να μπουν στην πρωτοπορία ή αν θέλετε να μπουν ενεργά στην ε, ευφυή εξειδίκευση. Όλη η επιτυχία ε, νομίζω βασίζεται καταρχήν στη διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που μπορούν να δώσουν έμφαση στην καινοτομία. Δηλαδή περιφερειακές αρχές, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κοινωνικοί φορείς. Νομίζω όμως ότι ιδιαίτερα οι περιφέρειες που έχουν αυτή την ανάγκη είναι και οι λιγότερο εξοικειωμένες με μια τέτοια συστηματική συνεργασία. Και αντιστοίχως, ενώ χρειάζεται καινοτομία και πολιτικά εργαλεία που θα ενισχύσουν την καινοτομία, αυτές οι περιφέρειες που έχουν σήμερα τα προβλήματα χαρακτηρίζονται και από έλλειψη πολιτικών για καινοτομία, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Το κρίσιμο λοιπόν είναι αφενός σε κάθε περιφέρεια να ενισχυθεί αυτή η αντίληψη ότι υπάρχει η ανάγκη συνεργασίας για μια προσέγγιση από τα κάτω προς τα πάνω έτσι ώστε σε κάθε περιφέρεια να εντοπιστούν τα δυνατά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες καινοτομίας και και απ' την άλλη η κάθε περιφέρεια ή οι περιφέρειες να συνεργαστούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδιαίτερα με εκείνες τις περιφέρειες που έχουν μεγάλη εμπειρία και τεχνοσία και έχουν μακριά παράδοση ακριβώς σε αυτούς τους τομείς. Τώρα, ε, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί νομίζω ότι επειδή είμαι και περιφερειακός σύμβουλος ε, και έχω μιλήσει με αρκετέ περιφέρειες υπάρχει μια έλλειψη κατανόησης στο τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δηλαδή νομίζω ότι το θέμα αυτό της ευφυού εξειδίκευση επικεντρώνεται κυρίως στην ανάθεση κάποιας μελέτης και κάποιος φορέας να προτείνει ιδέες για την καινοτομία. Δεν έχει κατανοηθεί δηλαδή ότι ο στόχος της ευθυούς εξειδίκευσης είναι απλώς κάποιος από τα πάνω ή κάποια εταιρεία να έρθει να προτείνει κάποιους τομείς αλλά αυτό να προκύψει ως διαδικασία συστηματικής διαβούλευσης, δημιουργίας δομών και μια σε βάθος ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιφέρειας. Και εκεί νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή αν οι περιφέρειες δεν κατανοήσουν τι σημαίνει ακριβώς ευφυής εξειδίκευση ε, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα και θα ανοίξει ψαλίδα μεταξύ περιφερειών που έχουν ήδη μια μεγάλη παράδοση και περιφερειών που θέλοντας να μπουν γρήγορα στην, ε, στην απορρόφηση πόρων του επόμενη της επόμενης προγραμματικής περίοδου θα κάνουν κάποιες, κάποιους πρόχειρους σχεδιασμούς. Ε, εκεί νομίζω πρέπει να βοηθήσουμε λίγο ίσως στην ενημέρωση και η Κομισιόν ίσως και εμείς ως Κοινοβούλιο να βοηθήσουμε λίγο στην ενημέρωση. Θα πρότεινα καταρχή εάν μπορούμε να οργανώσουμε μια ημερίδα στο κοινοβούλιο και να προσκαλέσουμε ακριβώς εκείνες τις περιφέρειες που έχουν λιγότερη εμπειρία και λιγότερη τεχνοσία πάνω στο θέμα της εξειδίκευσης. Αυτό θα τις βοηθήσει να κατανοήσουν σε ένα επίπεδο πιο οικείο το τι πρέπει να κάνουν. Το δεύτερο είναι προφανώς να ενθαρρύνουμε και τους κοινωνικούς εταίρους σε κάθε περιφέρεια, βέβαια δεν μπορούμε να φτάσουμε σε όλους, αλλά ίσως μέσα από ευρωπαϊκά δίκτυα να ενημερώσουμε λίγο για τη στρατηγική της ευθύους εξειδίκευσης ώστε όχι μόνο οι περιφέρειες αλλά αντιστοίχω και οι άλλοι κοινωνικοί φορείς είτε αυτοί είναι δίκτυα περιβαλλοντικών οργανώσεων είτε δίκτυα κοινωνικών φορέων είτε δίκτυα πανεπιστημίων ε, είτε δίκτυα μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κάθε, μέσα από ομοσπονδίες να κινητοποιήσουμε λίγο περισσότερο αυτούς του φορείς ώστε να μεταφέρουν τα μηνύματα ε, σε κάθε περιφέρεια. Και χρειάζεται νομίζω επίσης ενισχυμένη βοήθεια τεχνική προς τις περιφέρειες, ιδιαίτερα αυτές που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία. Ξέρω ότι η Κομισιόν έχει ε, χρηματοδοτεί και η Ρέτζιο χρηματοδοτεί κάποιους επιστήμονες και ειδικού για να βοηθήσουν τις περιφέρειες. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έχουν πλήρη γνώση και ενημέρωση περιφέρειες γι' αυτό και έχουν αξιοποιήσει αυτή τη ε, διαθεσιμότητα ειδικών για να βοηθήσουν. Και τέλος, νομίζω ότι δύο πράγματα επίσης είναι πολύ σημαντικά. Πώς θα εμπλέξουμε περισσότερους νέους σε αυτή τη διαδικασία σε περιφερειακό επίπεδο που ενώ έχουν γνώσεις και εμπειρία και τεχνοσία, από την άλλη μεριά είναι στο περιθώριο της διαμόρφωσης εξελίξεων, δεν συνδιαμορφώνουν τι εξελίξει, αυτοί οι άνθρωποι πώ θα μπουν στη διαδικασία να συνδιαμορφώσουν εξελίξει και δεύτερο, μερικέ θεματικέ ενότητε προτεραιότητα πρέπει επίση να είναι στο τραπέζι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, όπω είναι η οικονομία χαμηλού άνθρακα, η ε, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η αποτροπή των κινδύνων που συνεπάγεται, τα θέματα τη αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων, οι βιώσιμε μεταφορέ και όλα αυτά τα σχετικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Κορνέλια. Äh, Για να είμαι σύντομη. Είναι καλή η έκθεση, αν και είναι δύσκολο να αντιληφθούμε την ε, έξυπνη εξειδίκευση. Και εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει, αλλά κάπου είχε ε, οριστεί και από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτό τον όρο. Εν πάση περιπτώσει τώρα, επί της ουσίας, ε, σημαντικό είναι το θέμα της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών. Πρέπει να σκεφτούμε κάποιες πλατφόρμες, ε, την Επιτροπή των Περιφερειών, τη θεσμοποίηση της συνεργασίας. Αλλιώς υπάρχει μια τάση ε, κάποιων ε, ημερίδων ε, με τελείως προαιρετικό χαρακτήρα. Είναι λοιπόν σημαντική ιδιαίτερα η εξωτερική διάσταση επίσης. Τώρα, για την καινοτομία ήδη ακούστηκε για τον ορισμό της καινοτομία πως υπάρχει κοινωνική καινοτομία, όχι μόνο τεχνολογική, οικολογική καινοτομία ε, για να ξεκαθαρίσουμε πως δεν μιλάμε μόνο για τεχνολογικές ε, διαδικασίες. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για αυτό το οποίο λέτε σύγχρονη νοοτροπία των αρχών. Ε, είναι σοβαρό το ζήτημα της γραφειοκρατίας. Τώρα, δεν ξέρω αν ε, στέκουν όλα αυτά που αναφέρουν μας, αλλά είναι, είναι ένα ζήτημα πράγματι που έπρεπε να τεθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος τον λόγο. Πριν δώσω το λόγο στον Μιγγέλ να ρωτήσω κάτι άλλο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για τα μελλοντικά σχέδια της Κομισιόν σε σχέση με την πλατφόρμα της Σεβίλης, ε, Τι θα γίνει στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές και τι βλέπετε και πώς θα εμπλακούν οι υπόλοιπες ε, ευρωπαϊκές περιφέρειες στην πλατφόρμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σαν μια πρώτη, αν θέλετε, άμεση αντίδραση, η έκθεση είναι καλή και κυρίως είναι χρήσιμη. Και είναι χρήσιμη γιατί είναι εύθετη χρονικά. Λοιπόν, τρία είναι τα βασικά σημεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Το πρώτο αφορά τις νέες μεθόδους διακυβέρνησης και τις προτεραιότητες στις οποίες αναφέρθηκαν και κάποια μέλη σας. Εμείς θεωρούμε ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μια επίσημη τυπική υποχρέωση. Όπως λέτε εσείς πρόκειται για κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι ε, νομικά δεσμευτικό. Όχι, εμείς θέλουμε μια δυναμική διαδικασία, πειραματική διαδικασία, μακροπρόθεσμη διαδικασία που εμπλέκει κυρίως επιχειρήσεις και πανεπιστήμια. Σαν παράδειγμα, σήμερα βλέπουμε στην Πολωνία ότι για πρώτη φορά 500 επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί στην προγραμματική περίοδο των προγραμμάτων που θα ακολουθήσουν. Ε, έχουμε, έρθει, έχουμε κάνει 900 επαφές στην Κύπρο, έχουμε πάει στην Εστρεμαδούρα της Ισπανίας, έχουμε έρθει σε επαφή με μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθορίζοντας τις προτεραιότητές τους. Δεν μπορεί κανείς να επιβάλλει την, κοινότητα την καινοτομία. Μπορεί όμως να την καλλιεργήσει χωρίς να έχει μια αυστερά τεχνοκρατική αντίληψη. Να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ανοιχτής συμμετοχής με ελεύθερη καινοτομία. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο και έρχομαι στην τελευταία παρατήρηση. Μιλάμε για αιρεσιμότητα. Αν θέλει κανείς χρήματα την επόμενη φορά από το Περιφερειακό Ταμείο πρέπει να έχει μια σωστή στρατηγική. Και αυτό αποδίδει. Είδαμε ότι έχουν υπογραφεί μέχρι τώρα, ανεπίσημα βέβαια, έχουμε λάβει μάλλον μέχρι τώρα 13 εταιρικές τέτοιες συμφωνίες. Οι δυσκολίες που έχουν κάποια υπουργεία να επικοινωνούν είναι μια πραγματικότητα. Αλλά για πρώτη φορά βλέπουμε σε ορισμένες χώρες να γίνονται οι προσπάθειες το Υπουργείο που ασχολείται με την έρευνα, το Υπουργείο που ασχολείται με την οικονομία, το Υπουργείο που ασχολείται με την παιδεία έρχονται σε επαφή και συνεργάζονται. Αυτό γεννά την καινοτομία. Δεν μιλάμε μόνο για υψηλή τεχνολογία. Δεν μιλάμε για μια στενή ε, σχέση ανάπτυξης και έρευνας. Μιλάμε για καινοτομία με την ευρύτερη δυνατή έννοια. Και μιλάμε επίσης και για κοινωνικές καινοτομίες. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε και κάποιες κοινωνικές προκλήσεις που δυστυχώς υπάρχουν. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να δούμε τι ε, προσπαθούμε να κάνουμε με το ITTS. Έχουμε ήδη 13 κυβερνήσεις που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα αυτή και 139 περιφερειακές αρχές. Ε, ήδη καλύπτουμε τα τρία τέταρτα της ευρωπαϊκής γεωγραφίας. Η Ρουμανία και η Ιρλανδία ε, πλάκησαν τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε για μία πλατφόρμα που επιτρέπει και τον καθορισμό των στρατηγικών και την εφαρμογή των στρατηγικών. Δεν είναι εκ των άνω απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μέσω ανοιχτών δικτύων. Οι περιφερειακές αρχές αξιολογούν η μία την άλλη, συμβουλεύουν η μία την άλλη. Έχουμε 90 εμπειρογνώμονες που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθούν να βοηθήσουν αυτούς που το επιθυμούν. Προσπαθούμε να διευρύνουμε την πλατφόρμα αυτή κατά τη διάρκεια των επομένων ε, τριών ετών, έχοντας τις απαιτούμενους ελπίζουμε πόρους. Και προετοιμάζουμε και τα πιλωτικά προγράμματα, τα οποία έχουν καταθέσει και ο κύριος Βανίστελ Ρόι και το πιλωτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα σε μία από τις πιο φτωχές ε, περιοχές της Ελλάδας. Τώρα, οι, διαπα... οι διαπεριφερειακές συνέργειες. Πρώτον, οι συνάδελφοι στη Σεβίλη χαρτογραφούν για πρώτη φορά τις εξειδικεύσεις των περιοχών παράλληλα με τα πεδία αρμοδιότητας και τα ενδιαφέροντα των άλλων περιοχών για να μπορέσουν να έλθουν σε καλύτερη επικοινωνία. Η χαρτογράφηση δεν αρκεί, αν και κάνουμε βέβαια κάποια ειδική προσπάθεια στις νέες τεχνολογίες. Έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα έτσι ώστε οι περιφέρειες να μπορούν να δαπανίσουν το 15% ενός λειτουργικού προγράμματος για την καινοτομία σε άλλη χώρα. Οπότε έτσι διευκολύνουμε την διαπεριφερειακή συνεργασία. Εργαζόμαστε επίσης και στα πλαίσια του νέου Interreg για να μπορέσουμε να στηρίξουμε ε, τις συνεργασίες ανάμεσα στις ομάδες ε, των επιχειρήσεων και των πυρήνων, τα clusters τα λεγόμενα. Σας ευχαριστούμε επίσης γιατί στις 8 Νοεμβρίου αποφασίσατε να φιλοξενήσετε και αυτό ανταποκρίνεται και σε αυτά που είπε και ο συνάδελφος από την Ελλάδα, μια σημαντική πολιτική συνάντηση στην οποία θα είστε εσείς πρόεδρε, ο κύριος Βαν οι δύο επίτροποι, τρεις γενικοί διευθυντές. 400 έχουν καταγραφεί, εγγραφεί ε, για να πάρουν μέρος στην ακρόαση αυτή και θα είναι μια καλή ε, ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτήν την ε, ευφυή, εν πάση περιπτώσει, μορφή συνεργασίας. Ελπίζουμε επίσης να υπάρξει συνέργεια ανάμεσα στα διαρθρωτικά ταμεία και ε, στο, ε, στη στρατηγική 2020 μέχρι τις αρχές του Δεκεμβρίου. Δεν ξέρω, ε, δεν υπάρχει άλλο σχόλιο λοιπόν. Να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 18η Οκτωβρίου, την επόμενη Παρασκευή δηλαδή, 12η μεσημβρινή. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνάδελφοι, κλείνουμε το θέμα αυτό και τώρα θα περάσουμε αμέσως στις ψηφοφορίες. Ενθυμίστε ότι είχαμε υιοθετήσει μια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη, συνεπώς δεν θα ψηφίσουμε τα θέματα 5 και 6, οπότε ψηφίζουμε το 7, την έκθεση του κυρίου Τυρολιά Ελέγξτε παρακαλώ πρώτα εάν λειτουργούν οι κάρτες σας. Ελέγχουμε το μηχάνημα. Λίγοι ψήφισαν στη δοκιμαστική ψήφο. We have μείνετε παρακαλώ μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας γιατί δεν είμαστε και πάρα πολύ. Καλώς λοιπόν, όπως σας είπα θα ψηφίσουμε την έκθεση του Τυρολιά. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή πρώτα. Yeah, you go out, uh, Monsieur Κύριε Τυρολιά, θέλετε το λόγο. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς της νήσου Μαγιώτου τροποποιήθηκε στις 12 Ιουλίου του 12 από την 1η Ιανουαρίου του 14. Από την 1η Ιανουαρίου του 14 το αρχιτελ, αρχιπέλαγος της Μαγιώτ μετατρέπεται σε υπερπεριφερική ζώνη σύμφωνα με το άρθρο 355 της συνθήκης το κοινοτικό δίκαιο θα εφαρμοστεί στην Μαγιώτα από την 1η Ιουλίου του 2014. Θα υπάρξουν συγκεκριμένα προγράμματα και η εφαρμογή τους εξαρτάται από την ικανότητα της νήσου να σεβαστεί την κοινοτική νομοθεσία σε σχέση με τις υποδομές. Λόγω ακριβώς των περιορισμών της περιοχής αυτής έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιες εξαιρέσεις και κάποιες νομικές ρυθμίσεις έτσι ώστε να υπάρξει μια σταδιακή μετάβαση προς το κοινοτικό κεκτημένο. Καλούμεθα να ψηφίσουμε σήμερα δύο νομικές εκθέσεις, νομοθετικές μάλλον προτάσεις, για την μαγιότητα στον τομέα της αλληγίας και της ποιότητας των υδάτων στην Ίσο πρέπει ε, να ακολουθήσουμε τρεις ε, κατευθύνσεις θα έλεγα. Πρώτον, ισότητα ανάμεσα σε όλες τις περιοχές, όλες οι χώροι εξαιρέσεων και παρατάσεων μεταβατικών. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε μια νομική ασφάλεια και ικανοποιητική για τα εδάφη αυτά. Οι εξαιρέσεις αυτές προστατεύουν την Γαλλία από κάθε καταχρηστικές προσφυγές ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όπως γνωρίζετε η εφαρμογή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων εντάσσεται σε ένα πλαίσιο αιρεσιμότητας το οποίο μπορεί να δημιουργήσει θέματα στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που τόσον χρειάζεται η νήσος Μαγιότ. Όλες οι υπόλοιπες άλλες ε, περιφέρειες ε, ε, δυστυχώς έχουν τα ίδια προβλήματα τα οποία καθιστούν κάποιες ρυθμίσεις ευρωπαϊκές μη εφαρμόσιμες στην περιοχή. Σαν παράδειγμα έχουμε το πρόβλημα με την αλληλεία λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό, χωρίς βέβαια να προκαλέσουμε προβλήματα στην ενιαία αγορά όλα αυτά τα τοπικά θέματα και τοπικά προβλήματα με κάνουν να επανέλθω στο 349 της συνθήκης και να το εντάξω στη νομική βάση της ρύθμισης. Και να πω ότι έχω κουραστεί λίγο από την αιμονή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αρνείται επανειλημμένα την χρήση του 349 ως νομικής βάσεως της πρότασής μας, γιατί είναι κάτι το οποίο άπτεται του κοινοτικού δικαίου που εφαρμόζεται στην Ίσο Μαγιότ. Όλα αυτά είναι εγγεγραμμένα στη συνθήκη και προβλέπεται από ό,τι νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λειτουργήσει σαν θεματοφύλακάς της. Κάποιες άλλες τροπολογίες προτείνουν μια πιο ουσιαστική ε, χρονική αν θέλετε πρόβλεψη για την εξυγίανση των υδάτων της περιοχής. 200 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της επόμενης δημοσιονομικής περίοδου επί τη βάση κριτηρίων αφαίρετων μερικές φορές. Γι' αυτό λοιπόν οι πραγματικές ανάγκες φτάνουν τα 600 εκατομμύρια ευρώ και αυτό δείχνει ότι η Ευρώπη δυστυχώς φιλοδοξίες έχει αλλά δεν διαθέτει τα μέσα να τις εξυπηρετήσει τίθεται επίσης και το θέμα γενικότερα της ιδιοκτησίας στην περιοχή που καθιστά τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφικτες. Στην Αλία έχουμε την κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Εδώ δίδεται η δυνατότητα στην παράκτη Αλία να αναπτυχθεί στη Μαγιότ, σεβόμενη τα ανώτατα όρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της Υποεπιτροπής για τον Ινδικό Ωκεανό. Ξέρετε ότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο, πρέπει αυτά να λειτουργήσουν την 1η Ιανουαρίου του 2014. Η Πρόεδρος επιτάχυνε την διαδικασία έτσι ώστε η Αλληλεία, η Επιτροπή Αλληλείας και η δική μας Επιτροπή να γνωρίζουν ακριβώς ποια είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που θα συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό των σκέψεών μας μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Να σας εξηγήσω ότι δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο μέχρι σήμερα να συνδυάσουμε την προσπάθεια με την Επιτροπή Αλληλείας και να ακολουθήσουμε την τρέχουσα διαδικασία. Και αυτό δημιούργησε προβλήματα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ψηφίσουμε τις εκθέσεις αυτές σήμερα. Έγιναν όλα κάπως γρήγορα, αλλά καταλήξαμε στο να ψηφίσουμε σήμερα. Δεν μπορούσαμε όμως δυστυχώς να είχαμε προηγούμενες συζητήσεις. Λοιπόν θα ψηφίσουμε την τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Αποχές δεκτή, 4 υπέρ. Κατά, κατά. αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε γιατί δεν, σηκώνω δεν τα χέρια οι Ευρωπαϊκή Δημοκράτηση. λοιπόν θα επαληθεύσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 12 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στα εκτιμώντα. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 9 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Στα εκτιμώντα. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά να επαληθεύσουμε τη 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας δεκτή. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας εγκρίνεται 25 έναντι 4 έναντι μίας ψήφου και 4 αποχών περνάμε στην επόμενη γνωμοδότηση Τυρολιάν περνάμε στην ψηφοφορία το σημείο 8 της ημερικής διάταξης θα ήθελα να ξεκινήσουμε το 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20, 12 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή εκτιμώντας 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 3 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 16 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 4 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. 27 υπέρ, 4 αποχές εγκρίνεται. Περνάμε σημείο 9. Ρώσα Εσταράς Φερεγκούτ. Το σημείο 9. Uh, ε, can start the vote? Amendment 2 in favor. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 14 υπέρ, κατά να επαληθεύσουμε το 14, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία άρχεται πέρας απορρίπτεται περνάμε σε 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό, μέρος δεύτερο υπέρ, κατά αποχές δεκτό, 19 υπέρ, 19 υπέρ, να το επαληθεύσουμε, τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, 26 και 5 ψήφοι κατά. Η 20 υπέρ, Συγγνώμη Λαμπέρ. Δεν δε σε ακολουθούν από πίσω. Ε, δεν ξέρω ποιος κάνει κομμάτι στην ομάδα σας. Ο Τζέλερ. 20 υπέρ και πάλι. Κατά αποχές δεκτή. 21 με προφορική τροπολογία. Είναι κάποιος κατά της προφορικής τροπολογίας. Όχι. 21 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 4, επίσημη προφορική τροπολογία. Είναι κάποιο κατά, όχι, όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά αποχέ, δεκτή. 22 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ, κατά αποχέ, δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ, κατά αποχέ, δεκτό. Τροπολογία 5 υπέρ. Να επαληθεύσουμε το 5. Πέρας. Εγκρίνεται. 18, 13, 6 υπέρ. Κατά. Να το επαληθεύσουμε και αυτό, δεν είναι σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 27 δεν είναι συμβατή ε, με την ορθή πρακτική. Λοιπόν, εκτιμώντας 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 1 υπέρ. Να υπολυθεύσουμε την τροπολογία 1, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας δεκτή. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 9 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 10 προφορική τροπολογία, κάποιος κατά, όχι, ψηφίζουμε, όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Να την επαληθεύσουμε. Πέρας, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά Επαληθεύουμε την 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 17 με 12. Εκτιμώντας 12 υπέρ. Κατά... Α, και πάλι τα ίδια. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Την τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. And it is adopted 29 to 1. Εγκρίνεται με μία αποχή. Σημείο 10. Μαρή Τερέζη Σάντσε Σμιτ. Um, amendment. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ να ε, κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση στο 3 άρχεται η ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται 19 υπέρ 12 κατά τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ επαλήθευση για το 5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 Κανένας δεν ε, ε, σήκωσε το χέρι του. Ναι, ε, εσύ μόνο σου όμως, κανένας άλλος. Εντάξει, επαλήθευση, δεν σε ακολούθησε κανείς. επαλήθευση για το 12. Πέρας. Και απορρίπτεται. 13 υπέρ, 18 κατά. Τροπολογία 61 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ Κατά. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά δεν είμαι βεβαία. Επομένως, επαλήθευση. Τροπολογία 13. Πέρας. Απορρίπτεται 14 υπέρ 17 κατά. Τροπολογία 62. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Ε, επαλήθευση για τη 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 18 υπέρ, 15 κατά. Τροπολογία 17 υπέρ. Ίδια κατάσταση, επαλήθευση επί της 17, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 17 υπέρ 15 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 18 υπέρ 15 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ επαλήθευση για 19 άρχεται. Πέρας. 17-15 εγκρίνεται. Τροπολογία 20, επαλήθευση επί της 20. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ κοντινό, εν πάση περιπτώσει. Πέρα στις ψηφοφορίες 17 υπέρ, 15 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Ίδια κατάσταση. Θέλετε να επαληθεύσουμε ή να θεωρήσουμε ότι είναι ίδιο αποτέλεσμα. Όχι, ελέγχουμε. Πέρας της ψηφοφορίας 17-15 εγκρίνεται τροπολογία 22 ίδια κατάσταση. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 17-15 εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Ε, για την τροπολογία 23 παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 18 προς 15 εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 27. Επαλήθευση για την τροπολογία 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 28 υπέρ κατά επαλήθευση για την 28 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 19 προς 12 εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 επαλήθευση. Επαλήθευση της τροπολογίες 29. Πέρας. 17 ε, προς 16 εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Επαλήθευση και για την τροπολογία 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 20 προς 13, 31, Τρία τροπολογία 31, υπέρ, όχι, ελέγχουμε, Η ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 17 προς 16, 32 υπέρ, κατά. Ναι, ε, συνέχεια θα είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, τι θέλετε, ε, μου έχετε εμπιστοσύνη, τεκμέρουμε ότι, είναι, ε, ότι εγκρίνεται. Ναι, αλλά μπορεί κάποια φορά το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό. Λοιπόν, 32 έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 32. Νομίζω η ίδια... Ε, Α, όχι, 20 υπέρ, 13 κατά, ναι. Επομένω και εδώ η ηλεκτρονική επαλήθευση, πέρασε τέλος, ίδιο 18 υπέρ 13 κατά 3, τροπολογία 68, όχι, καταπίπτει, 69 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται, 14 υπέρ, υπέρ, επαλήθευση, δεν καταλαβαίνω το αποτέλεσμα. closed. Πέρα τη ψηφοφορία απορρίπτεται 14 υπέρ 15 κατά. Βλέπετε ότι είχα δίκιο, πρέπει να επαληθεύουμε. Λοιπόν, 70 υπέρ κατά απορρίπτεται, 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τι θέλετε. 72 πάμε, υπέρ. Η 71 απερίφθη. Άρα ψηφίζουμε την 34, τροπολογία 34 υπέρ. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 34 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 15 υπέρ, 15 κατά απορρίπτεται. Κάποιος παρακοιμήθηκε και δεν ψήφισε. 72 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 35. 35. Λαμπέρ, το χέρι σου. Ηλεκτρονική επαλήθευση πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνει τα 17 υπέρ 13 ε, κατά. Τροπολογία 36. 36. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37. Λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 37. Εγκρίνεται 16 υπέρ 14 κατά. Τώρα πάμε στην τροπολογία 73 υπέρ. Λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 73, άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 16 υπέρ, 14 κατά, επομένως δεν θα ψηφίσουμε την 40. Πάμε τροπολογία 41 υπέρ, υπέρ της 41. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42-74 ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ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 αν θέλετε, μπορούμε να πάμε και λίγο πιο πίσω. Ποια τροπολογία θέλετε, σε ποια θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. 49, 49 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 52, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 18 υπέρ 13 κατά εγκρίνεται, 53 υπέρ επαλήθευση μάλλον και για την τροπολογία 53, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 18 προς 13 εγκρίνεται, 54 υπέρ ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 54, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 18 υπέρ 13 κατά εγκρίνεται, 55 υπέρ επαλήθευση από τις 55 Πέρας. 18 υπέρ, 13 κατά εγκρίνεται τροπολογία, 56 υπέρ, ίδια κατάσταση μάλλον. Πιστεύω ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται 18 προς 13, 57 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 58 υπέρ. «58 εγκρίνεται». Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία αυτή τη φορά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Σημείο 11 της ημερησίας διατάξεως. Ιωαχήμ Τσέλερ, γνωμοδότηση Ιωαχήμ Τσέλερ. Τροπολογία 24, τροπολογία 24 λέω υπέρ κατά. Όλοι είναι κατά, επομένως απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται ε, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 1 άρχεται πέρας και απορρίπτεται 14 ψήφι υπέρ 18 κατά τροπολογία 2 υπέρ Ηλεκτρονική επαλήθευση η τροπολογία 2. Ενδεχομένως θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 16 υπέρ 15 κατά. Ένας δεν ψήφισε, δεν ξέρουμε από ποια πλευρά. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 3 άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται 17 προς 15. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται 17 προς 15. Τροπολογία 35 υπέρ. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 35. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 17 προς 15. Τροπολογία 36, ενδεχομένως το ίδιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση και για την τροπολογία 36. Πέρας της ψηφοφορίας. Και 16 προς 15 εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13,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 υπέρ αποχές απορρίπτεται. 45 δεν είναι συμβατή με την ε, σωστή ε, νομοθετική διατύπωση. Μ' αρέσει αυτό, η αυτή η διατύπωση. Λέει 14 υπέρ αποχές απορρίπτεται, 15 υπέρ αποχές απορρίπτεται, 16 υπέρ αποχές απορρίπτεται, 17 υπέρ αποχές απορρίπτεται, 18 υπερκατά αποχές απορρίπτεται, 19 υπερκατά αποχές απορρίπτεται, 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 21 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση από τις τροπολογίες 29. Ευχαριστώ Κωνσταντς, γιατί είχα αρχίσει να βαριέμαι με αυτό το υπέρ κατά. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας 17 υπέρ 15 κατά, επομένως εγκρίνεται τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές, ίδια κατάσταση, ηλεκτρονική επαλήθευση επομένως. Τροπολογία 22, ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. 17 υπέρ 15 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 23, η ίδια κατάσταση. Όχι, απορρίπτεται βλέπω, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν, άρχεται. Πέρας. 29 υπέρ, καμία ψήφος κατά τρεις αποχές. Επομένω ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Περνάμε στην γνωμοδότηση του Fris Βλάσακ σχετικά με το περιφερειακό σήμα ποιότητας. Συμβιβασμό 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Η ηλεκτρονική επαλήθευση τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 12 υπέρ 20 κατά. Ε, συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά υπέρ υπέρ. Όχι. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 12. Πέρας. 17 υπέρ 14 κατά εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 16. Πέρας της ψηφοφορίας 17 υπέρ 15 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά. Τροπολογία 19 λοιπόν. 19 υπέρ. Όχι, θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση, δεν είμαι βεβαία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη 13 προς, 20. Η 20, ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη 13 προς 19. Συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ η ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 26. Πέρας και απερίφθη 13 προς 18 με μία αποχή 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 28 έχει αποσυρθεί 30, ναι, ψηφίζουμε την 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 Ποια τροπολογία ψηφίζουμε τώρα λέει η Πρόεδρος Ψηφίζουμε την 29 Εγκρίναμε την τροπολογία 28 Ψηφίζουμε την 29 υπέρ. Τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 29. Πέρας. Απερίφθη 14 προς 18. Και έχουμε τώρα την τροπολογία 31 υπέρ. Θα κάνουμε και εδώ ηλεκτρονική επαλήθευση καλύτερα. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν για την τροπολογία 31. Πέρας της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται 17 υπέρ 14 κατά ε, ηλεκτρονική τελική ψήφος. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία πέρας. Το αποτέλεσμα 30 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, συγχαρητήρια. Και περνάμε τώρα στο σημείο 13. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε περίπου μία ώρα στη διάθεσή μας. Έχουμε μία γνωμοδότηση και δύο εκθέσεις. We most likely we might not make the, uh, the, last point. Το τελευταίο σημείο ίσως να μην το προλάβουμε. Ελίζαμπετ, θέλετε να αναβάλουμε το τελευταίο θέμα την επόμενη φορά ή να ξοδέψουμε 20 λεπτά μόνο για κάθε έκθεση και γνωμοδότηση. Αν κάνουμε κανονικά τη διαδικασία το τελευταίο σημείο δεν θα το προλάβουμε. Ή θα συμφωνήσουμε 20 λεπτά για κάθε έκθεση ή η δική σου έκθεση πάει τον Νοέμβριο. Οι συντονιστές θα πρέπει να το αποφασίσουν αυτό. Μπορούμε να την αναβάλουμε αν θέλετε. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι πρέπει να την αναβάλουμε. Ήδη το έχουμε κάνει. Δεν ξέρω αν μπορούμε μια άλλη έκθεση να μετακινήσουμε. Δεν ξέρω σε τι θα χρησιμεύσει εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η ιστορία. Από την άλλη έχω καταθέσει το κεντρικό ε, έγγραφο, έχω ήδη συλλέξει αντιδράσεις, και όσοι ε, θέλουν να κάνουν παρατηρήσεις μπορεί να τις κάνουν και γραφτά συνάδελφοι. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν το πιο σωστό. Αυτή κανονικά θα έπρεπε να είναι η πρώτη συζήτηση έτσι και αλλιώς. Να έρθετε σε επαφή μαζί με την Μπεθ λοιπόν έτσι ώστε να αντιστείλετε τα σχόλιά σας. Θα ξεκινήσουμε τώρα με την έκθεση Κάντενμπαχ. Φιλόξενο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Έχουμε και δύο σκιώδεις που θα πάρουν το λόγο, γι' αυτό παρακαλώ να είστε όσο πιο σύντομοι γίνεται. Κυρία Κάντενμπαχ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Σε καιρούς τέτοιους πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε κατά νου πως η πολιτική συνοχή είναι σημαντικό μέσο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Πρέπει αυτό να το έχουμε πάντα κατά νου και υπάρχουν πολλές δυνατότητες να εκμεταλλευτούμε αυτό το δυναμικό που υπάρχει, ειδικά για να προωθήσουμε την απασχόληση των νέων. Θεωρώ πως ε, υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την ε, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ειδικά σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν δούμε πως ε, αυτές δημιουργούν τις περισσότερες ε, θέσεις εργασίας και μην ξεχνάμε πως αν έπαιρνε κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις ένα παραπάνω εργαζόμενο θα είχαμε καταπολεμήσει την ανεργία στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία του Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και του Επενδυτικών Ταμείων για να βοηθήσουμε την ίδρυση νέων τέτοιων επιχειρήσεων. Και βεβαίως και ο Τζοζεφ Στίγκλιτς, ε, νομπελίστας, είχε πει πως ε, οι επιχειρήσεις ιδρύονται εκεί όπου υπάρχει εμπιστοσύνη ε, και μπορούν να βασιστούν γιατί μόνο έτσι μπορεί να ανθίσει η επιχειρηματικότητα. Και νομίζω αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου ειδικά σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, εάν κάτι πάει στραβά και αποτύχει η επιχείρηση, πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική ε, διασφάλιση. Χρειαζόμαστε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και από πλευράς ε, υγείας, μια ισορροπία μεταξύ οικονομικών ε, και κοινωνικών πτυχών. Ακριβώς ε, για να υπάρχει η δυνατότητα προώθησης επιχειρηματικότητας, για να ιδρύονται επιχειρήσεις και να δημιουργεί ένα περιβάλλον εντός του οποίου θα δραστηριοποιούνται οι ε, επιχειρηματίες. Επίσης, χρειαζόμαστε ασφαλείς και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας ε, γιατί βεβαίως δεν είναι δυνατόν οι επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους δεν είναι αυτή η Ευρώπη την οποία φανταζόμαστε. Επίσης θα ήθελα να πω να, πως πρέπει να αναφέρουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Υπάρχουν ε, πολλές ε, βέλτιστες πρακτικές, δεν χρειάζεται να αφευρίσκουμε κάθε φορά τον ε, τροχό πρέπει να δούμε τα μοντέλα τα οποία έχουν ήδη αποδειχτεί αποτελεσματικά. Πρέπει λοιπόν ε, τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες να παρουσιάσουν αυτά τα επιτυχή μοντέλα, να μάθουν ε, ο ένας από τον άλλον και ένα άλλο πρόβλημα που ακούμε συνεχώς όταν μιλάμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Εδώ πέρα πρέπει να βρεθούν λύσεις που θα δίνουν την δυνατότητα πρώτον βεβαίω να ιδρυθούν επιχειρήσεις και δεύτερον να επεκταθούν για να είναι εύκολη και μη γραφειοκρατική η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Και βεβαίως ε, κάτι άλλο το οποίο λέμε παντού ότι πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία αλλά από την άλλη να υπάρχει και ασφάλεια για τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τα λεφτά του Ευρωπαίου φορολογούμενου και την διαφανή χρήση τους. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ, Λαμπέρτ Φανίστελ ε, Ναι, δεν ήξερα πως ε, θα ήμουν σκιώδης ηγητής. Αυτό το οποίο θέλω εγώ να πω είναι ως ο συνδυασμός με μια γενικότερη προσέγγιση και τα ευρωπαϊκά ταμεία επενδύσεων και τα διαρθρωτικά ταμεία σχετίζεται και με τις δυνατότητες ε, του διαδικτύου. Ε, ειδικά σε μέρη όπου δεν βρίσκεται κάποιος στο κέντρο, αλλά σε περιοχές της υπαίθρου ή σε μέρη που δεν είναι συνδεδεμένα με την ευρυζωνικότητα. Και τις μέρες αυτές υπάρχει μια έκθεση στο Κοινοβούλιο και μια συνάντηση με συμμετοχή της κυρίας Κρούση για την δυνατότητα που δίνουν οι δορυφόροι στις επικοινωνίες, ε, στην πλοήγηση πέραν των αστικών περιοχών. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό το οποίο επίσης είπατε είναι χρήσιμο δηλαδή να έχουμε νέες ε, μεθόδους που θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ε, στα διαρθρωτικά ταμεία και στα επενδυτικά ταμεία Ε, όπως οι επενδυτές ε, παραδείγματος χάρη που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις ε, ή να τους μάθουν τη χρήση του διαδικτύου. Και επίσης η μεγαλύτερη σχέση που πρέπει να αποκτηθεί με την χρηματοπιστωτική καινοτομία. Αυτές τις δύο προσαρμογές θα ήθελα να κάνω σημαντικό νομίζω. Επίσης πράγματι 95% των επιχειρήσεων είναι μικρές και μεσαίες. Οπότε για την αύξηση των θέσεων εργασίας έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις μεγάλες εταιρείες. Τέλος, πρέπει να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα κάποιας ε, εξειδίκευσης. Μιλήσαμε για έξυπνη εξειδίκευση και οι νέες αυτές επιχειρήσεις που ιδρύονται συχνά έχουν σχέση με το γενικότερο οικοσύστημα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μεγαλύτερων εταιριών ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή. Μία σχέση δηλαδή ε, μεταξύ νέων επιχειρήσεων ε, και του ευρύτερου περιβάλλοντος θα ήταν χρήσιμη. Σας ευχαριστώ κύριε Χρυσόγγελος. Ευχαριστώ πολύ είναι αλήθεια ότι η, κρίση πλήττει πολύ περισσότερο τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις γιατί δεν έχουν μεγάλη δυνατότητα προσαρμογής όσο πιθανά έχει μια μεγαλύτερη εταιρεία που έχει και αναπτυγμένες δομές. Ε, Απ' την άλλη μεριά, για να αντιμετωπίσουμε την κρίση δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε αποδόμηση του κοινωνικού προτύπου στην Ευρώπη. Δηλαδή να δουλεύουν οι άνθρωποι χωρίς να πληρώνονται στοιχειώδη μισθό, και ε, να αποδομήσουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το θέμα της έξυπνης εξειδίκευσης, αλλά αυτό πρέπει να αποτυπωθεί και στο πώς οργανώνονται οι επιχειρήσεις. Νομίζω ότι μέσα στην κρίση εμφανίζονται καινούργια μοντέλα οργάνωσης των επιχειρήσεων που περιορίζουν το κόστος μέσα από έξυπνες επιλογές, δηλαδή συνεργασία σε δίκτυα, όχι κατά ανάγκη ενοικίαση χώρων που ε, δημιουργούν ε, μεγάλο κόστο, στα πάγια κλπ. Ε, πρέπει να βρούμε λοιπόν και έξυπνου τρόπου χρηματοδότηση αυτών των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δεν θα περνούν κατά ανάγκη και μέσα από το τραπεζικό δρόμο ο οποίος απαιτεί συγκεκριμένε λειτουργίε, δηλαδή έδρα επαγγελματική, υποδομές κτλ. οι οποίες θα πιστοποιήσουν ότι μόνο αυτό το μοντέλο είναι βιώσιμο σε επιχείρηση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βρούμε ε, εργαλεία όπως είναι οι μικροχρηματοδοτήσεις. Δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Ε, μικροδάνεια, ε, συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που η μία μπορεί να δανείζει την άλλη και άλλα εργαλεία που θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά στο ξεκίνημα μικρών επιχειρήσεων που δεν χρειάζονται τεράστια κεφάλαια αλλά πολλές φορές χρειάζονται μικρά κεφάλαια για να μπορέσουν να ξεκινήσουν που όμως αυτά τα μικρά κεφάλαια δεν είναι εύκολο να τα βρούνε από το συστημικό τραπεζικό σύστημα και γι' αυτό νομίζω θα πρέπει και όλη η συζήτηση και για τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά και οι πρωτοβουλίες της να λαμβάνουν υπόψη και ένα εναλλακτικό μοντέλο μικρών χρηματοδοτήσεων. Ε, είναι αλήθεια επίσης ότι ο ρόλος των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί μπορεί να συνδυάσει επιχειρηματικότητα με κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος. Οπότε θα πρέπει να άρουμε εμπόδια τα οποία ε, εμποδίζουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα και σε δυνατότητες χρηματοδότησης η προηγούμενη περίοδο, για παράδειγμα στην Ελλάδα δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης ε, κοινωνικών επιχειρήσεων ή ακόμα και μη κυβερνητικών οργανώσεων σε προγράμματα μέσα από το ΕΣΠΑ, μέσα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί έτσι ώστε να μην δημιουργούνται υπερβολικά εμπόδια σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Και προφανώς θέλουμε λιγότερη γραφειοκρατία και άρση δυσκολιών, αλλά βέβαια αυτό πρέπει να συνδυάζεται με διαφάνεια για να μην σπαταλιώνται πόροι και νομίζω και εκεί πρέπει να δώσουμε και να δώσουν τα κράτη-μέλη έμφαση μεγαλύτερη στα θέματα της αποτελεσματικότητας και της αξιόπιστης χρήσης των ευρωπαϊκών πόρων για να παράγεται αποτέλεσμα και ιδιαίτερα να δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω εάν ε, η Κομισιόν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο, θέλει να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Και να μας πείτε και ποιο είστε, Ροδρίγο Πεντούτσι από τη DG Enterprise και Industry. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, κυρία Πρόεδρε. Φυσικά, στην ε, νέα προγραμματική περίοδο θα έχουμε ε, θα έχουμε ευθυγράμμιση της περιφερειακής πολιτικής με την πολιτική 2020 και φυσικά ε, ο τρόπος που μας απασχολεί εδώ είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους ε, για να δουλέψουμε επί τόπου. Επίσης ε, θέλουμε και προτιθέμεθα να εστιάσουμε την προσοχή μας στις start-ups αλλά οπωσδήποτε θα ε, παίξει ρόλο και ε, η βοήθεια που θα δώσουμε, η διαρθρωτική βοήθεια ε, στις νέες και τις μικρές επιχειρήσεις. Ε, μια μικρή ανακοίνωση μπορώ να σας κάνω εδώ. Ε, του χρόνου η Κομισιόν ε, θα συνεργαστεί στη δικιά μας Γενική Διεύθυνση και τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο έτσι ώστε να προλάβουμε κατά κάποιο τρόπο την εργασία επιτόπου. Πρόεδρος, πρέπει να αποφασίσουμε πότε θα είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες 18 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι, Παρασκευή δηλαδή 12 το μεσημέρι. Θέλετε να προσθέσετε κάτι συνάδελφε μετά τη συζήτηση. Ε, αν θέλετε μπορείτε να πάρετε το λόγο φυσικά. Επί της αρχής ε, τίποτα ιδιαίτερο. Σας ευχαριστώ. Ε, όποιος ε, θέλει βεβαίως να πει και να προσθέσει κάτι μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μου έτσι μέχρι την Παρασκευή. Ο Σόν. Ναι, συγγνώμη, έπρεπε να το είχα πει πιο νερό ότι θέλω να πάρω το λόγο. Εν πάση περιπτώσει εδώ ε, θέλουμε να ξεπεράσουμε την οικονομική ε, κρίση, αλλά σίγουρα αυτό θα γίνει μόνο εάν ε, μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως και δύο ζητήματα τα οποία δεν λειτουργούν και δεν αναφέρονται εδώ καλά. Ας πούμε τα ε, προγράμματα τα οποία είναι διαθέσιμα ε, και τα οποία δεν γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι και οι δυνάμοι δικαιούχοι. Επομένως θα πρέπει να ε, δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στην επικοινωνία, να δουλέψουμε με τις υπηρεσίες επιτόπου. Δεύτερον, όσον αφορά την διαθέσιμη χρηματοδότηση, να είναι πιο εύκολη η χρηματοδότηση, ευκολότερη από ό,τι είναι τώρα επίσης θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να αποτυγχάνουν. Θέλω να πω ότι ε, ε, ε, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η πρώτη αποτυχία μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για κάτι καλύτερο, για μια επιτυχία αργότερα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα σημαντικό βήμα η αποτυχία, ένα σημαντικό βήμα προς την επιτυχία. Τέλος έγινε και μια αναφορά σε αυτό, ε, είναι ότι η δημιουργία της ευρυζωνικότητας ε, σε όλη την Ευρώπη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η πρόσβαση δηλαδή στην ευρυζωνικότητα ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι ταχείες συνδέσεις είναι οπωσδήποτε απαραίτητες για τη δημιουργία ε, επιχειρήσεων. Λοιπόν, 18 Οκτωβρίου είπαμε ότι είναι η προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών. Ελπίζω ότι και θα προλάβεις ε, να υποβάλεις τροπολογίε σου. Ολοκληρώνουμε λοιπόν, περνάμε στο σημείο 14 της ημερησία διατάξεως, έκθεση Ντέρεκ Vaughan. Σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Την τελευταία ε, συνάντησή μας, την τελευταία συνεδρίασή μας είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις ε, σχετικά με το θέμα αυτό. Είναι Δίασα πρωτοβουλίας ε, έκθεση και ε, θέλουμε, θελήσαμε εδώ να κάνουμε ένα έγγραφο το οποίο να ασχολείται και με τα, το πολιτευτές δημοσιονομικό πλαίσιο και με την πολιτική συνοχή, να δούμε ποια θα είναι η επίπτωση στις περιφέρειες των χωρών. Επομένως, εδώ η έκθεση ε, έχει αποσκοπεί μάλλον στο να δούμε ποια είναι, ποια είναι τα επιχειρησιακά προγράμματα και ποια, ε, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε προχωρήσει. Ε, επομένως, μας ενδιαφέρει να δουν και οι συνάδελφοι εάν είναι και ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο έχουν ενσωματώσει τις παρατηρήσεις που είχαν κάνει. Ε, η ε, συνοχή είναι οπωσδήποτε σημαντική έτσι ώστε να υπάρξει οικονομική ε, ανάκαμψη και επομένως είναι και πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια, με ποιο τρόπο δηλαδή μπορούν να, δημιουργηθούν νέες αιρεσιμότητες, νέες δυνατότητες εταιρικών, εμπορικών και επιχειρησιακών σχέσεων κτλ. Εγώ προσπάθησα να βγάλω κάποια πρώτα συμπεράσματα ε, και ε, προσπάθησα και επιτόπου να δουλέψω πολύ. Νομίζω λοιπόν ότι ε, υπάρχουν πολύ διαφορετικά στάδια προετοιμασίας στις διάφορες χώρες μέλη. Πρέπει να πω ότι οι πιο νέες χώρες μέλη ίσως είναι πιο προχωρη, σε πιο προχωρημένο στάδιο από τις πιο παλιές χώρες μέλη. Προσπάθησα να δώσω και κάποιες αιτιολογήσεις όσον αφορά ή επεξηγήσεις όσον αφορά τις διαφορές που υπάρχουν. Ε, ενδεχομένως οι διαφορές αυτές προκύπτουν από την ε, διαφορά χρηματοδότησης, από το διαφορετικό στάδιο προετοιμασίας, από κάποια ε, ήδη υπάρχοντα προγράμματα επιτόπου. Ε, εξαρτώνται επίσης από το κατά πόσον έχουν εμπλακεί στις διαδικασίες τοπικές περιφερειακές ε, αρχές κτλ. Υπάρχουν επίσης ε, χώρες ε, μέλη οι οποίες ε, θέλησαν να συμπεριληφθούν στην όλη συζήτηση και άλλοι φορείς όπως μη κυβερνητικέ οργανώσεις κτλ. Επομένως μέσα από την προσπάθεια συνέργειας όλων αυτών των οργανισμών ενδεχομένως προκύπτουν κάποιες καθυστερήσεις δεν είναι δυνατόν βεβαίως να ε, είναι προφανές ότι όταν καταφέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συνεννοηθούν τότε θα είναι πιο αποτελεσματικός ο τρόπος ε, ε, χρήσης των, ε, των κονδυλίων. Ναι, πολύ σημαντικό είναι να ε, ε, υπάρχει και σαφής ε, καταγραφή όλων των προτεραιοτήτων, την δυνατότητα άντλησης χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά ταμεία, την δυνατότητα συνέχισης χωρίς μεγάλες παύσεις προγραμμάτων από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και άλλα που ξεκινούν στην επόμενη. Ε, στο τέλος της έκθεσης ε, αναφέρω πράγματι ότι ε, σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν χώρες οι οποίες ακόμα αγωνίζονται λίγο να ξεκινήσουν ενώ άλλες είναι σε πιο προχωρημένο βαθμό προεργασίας. Η εταιρική σχέση μπορεί να δώσει λύση στο μέλλον σε αυτό το πρόβλημα. Όσον αφορά τα partnership agreements έχουν ήδη υποβληθεί οι περισσότερες, υπάρχουν ακόμα κάποιες τα δε επιχειρησιακά προγράμματα, ε, μερικά έχουν ήδη υποβληθεί τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο και η Κομισιόν περιμένει τώρα κάποια άλλα. Προσπάθησα να μην ε, κάνω συγκεκριμένες αναφορές ε, στην έκθεση. Όσον αφορά τα τελικά συμπεράσματα, νομίζω ότι γενικά η έκθεση είναι, έχει θετικό πρόσημο και αντλούνται κάποια διδάγματα και συμπεράσματα όσον αφορά τον τρόπο που εφαρμόζονται εφαρμόζεται η πολιτική συνοχή στις διάφορες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Το συζητήσαμε το θέμα αυτό και στην τελευταία συνάντηση και βλέπω ότι κάποιες από τις παρατηρήσεις μας ε, έγιναν δεκτές. Ως εκ τούτου η έκθεση είναι μια σωστά σταθμισμένη έκθεση. Ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. να μας πούν τι εντυπώσεις έχουν διαμορφώσει από τις προετοιμασίες των εταιρικών συμφωνιών Για την Ολλανδία σαν παράδειγμα βλέπω ότι στην περίοδο από το 2007 χάσαμε πάρα πολύ χρόνο. Μόνο μία συμφωνία είχε συμφωνηθεί τον μήνα Δεκέμβριο. Και αυτές οι καθυστερήσεις που σημειώνονται είναι κάτι το οποίο με απογοητεύει. Έχουμε κάποιες υποσχέσεις από το Συμβούλιο σχετικά με το πώς θα πρέπει να κινηθούμε από εδώ και πέρα και πώς θα πρέπει να προπαρασκευαστούμε σωστά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πίεση πλέον, δεν πρέπει να καθυστερήσουμε άλλο Δεν ξέρω, ίσως να είμαι υπεραισιόδοξος, θα ήθελα όμως κάποιες πληροφορίες από πλευράς της Επιτροπής. Ο κύριος Χρυσόγελος. Χωρίς μικρόφωνο και ο κύριος Χρυσόγελος και η Πρόεδρος, δεν ακούσαμε. Äh, äh δεν είμαι σίγουροι αν είναι σωστός ο τίτλος ότι μιλάμε για την ε, ικανότητα δεν είναι θέμα διάθεσης δηλαδή είναι θέμα πραγματικά το εάν ε, όντως μπορούν το θέμα είναι βεβαίως να δούμε αν μπορούμε να επιφέρουμε καμία ε, ουσιαστική αλλαγή. Ναι, εντάξει, να δούμε πού βρίσκονται τα κράτη-μέλη, οπωσδήποτε. Αυτό είναι χρήσιμο, αλλά τώρα έτσι όπως παρουσιάζεται, δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία με εκνευρίζουν, θα έλεγα. Δηλαδή, λέτε, το είναι ικανότητα των κρατών μελών να κάνουν το χ και το ψ. Ε, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πως έχουμε σοβαρά προβλήματα ε, στο να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για τον προϋπολογισμό και τους ε, όρους ε, που επιβάλλονται. Δηλαδή είναι σχεδόν ηρωνία το να μιλάμε μετά για ικανότητα των, ε, και ετοιμότητα των κρατών μελών. Εντάξει, κάποια πράγματα υπόθηκαν για τον προϋπολογισμό ότι δεν βοηθάει πάρα πολύ να καταπολεμήσει και να αντισταθμίσει τις διαφορές που υπάρχουν και τώρα να μιλάμε, όπως είπαμε, για ικανότητα και ατιμότητα δεν έχουν μεγάλη σχέση με αυτό το θέμα. Πρώτον. Δεύτερον, κάποια άλλα σημεία τώρα. Ναι, εντάξει, ωραία, απλοποίηση. Ναι, και εγώ θέλω να απλοποιήσω πολλά πράγματα στη ζωή μου. Έτσι και τα κράτη-μέλη. Το εάν τώρα αυτό που διαβάζουμε εδώ πέρα, αν έχει σχέση με το αντικείμενο, δεν είμαι πολύ σίγουρη. Στρατηγική 2020. Σας πενθυμίζω πως είχαμε ασκήσει κριτική εδώ, σε αυτή την αίθουσα. Ξαφνικά εξαφανίζονται όλα και η σχέση με την πολιτική συνοχή ε, αποκαθίσταται σαν να μην συνέβη τίποτα, με τρόπο που δεν μπορώ να αντιληφθώ. Ε, ετοιμότητα. Εντάξει, ναι, να το κάνουμε, αλλά πρέπει να πάμε στους λόγους έτσι, γιατί έχει η κατάσταση ως έχει. Αυτή είναι η διαπραγματευσή που γίνεται εδώ πέρα. Ε, ε, και αυτή επηρεάζει και εδώ μέσα και αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διοικητικές ικανότητε, πράγματι οι ικανότητε διοίκησης του κάθε κράτους μέλους διαφέρουν. Και όταν μιλάμε για στρατηγική κάποιων κρατών μελών, ε, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, ε, και εκεί πέρα στρατηγική που και δεν βοηθούσε πάντα. Και μετά έχω και ένα ερώτημα προς ε, τον εισηγητή για τα επιχειρησιακά προγράμματα. Για μένα το θέμα δεν είναι το να έχουμε ένα, δύο ή δεκαεφτά επιχειρησιακά προγράμματα, αλλά κατά πόσον είναι συμβατά, ποια ποιότητα έχουν. Οπότε η συζήτηση αυτή για τα επιχειρησιακά προγράμματα θεωρητικά εντάξει μπορεί να ε, έχει λογική αν το δει κανείς ε, από σκοπιά κεντρικού κράτους, αλλά σε ομοσπονδιακά κράτη όπως η Γερμανία και άλλα ομοσπονδιακά κράτη στην Ένωση δεν έχει νόημα. Οπότε... Εντάξει, η συζήτηση καλή είναι, αλλά δεν ξέρω αν επιτυχάνουμε κάποια ουσιαστική βοήθεια εδώ πέρα. Ε, θα προτείνουμε και κάποια καλύτερα επιχειρήματα, αυτό δούμε. Thank you. Vlasak. Vlasak. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση είναι σημαντική, είναι μια έκθεση η οποία θα μας ενημερώσει σωστά θα έλεγα και με χρήσιμο τρόπο για τις εξελίξεις σε ένα τόσο σημαντικό τομέα. Καλό θα ήταν πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει περισσότερα στοιχεία και περισσότερα δεδομένα για αντίστοιχες συμφωνίες εταιρικού τύπου. Θα θέλαμε να μάθουμε αν είναι χρήσιμες οι συμφωνίες, αν έχουν φανεί χρήσιμες για τους εταίρους, αν έχει διευκολυνθεί η συμμετοχή των ε, τοπικών αρχών και των δημοτικών αρχών και αν πράγματι έχει εφαρμοστεί η λεγόμενη ε, ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Ο κύριος Χρυσόγελος έχει το λόγο και μετά ο Βίκτορ. Ε, είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε ορισμένα στοιχεία από την Κομισιόν για να δούμε ποια είναι η πραγματική εικόνα σήμερα της προετοιμασίας και των περιφερειών και των εθνικών κρατών. Ε, νομίζω ότι δεν έχουμε αυτή την εικόνα. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ορισμένα σημεία στην έκθεση. Ε, και στην Επιτροπή εδώ αλλά και γενικότερα νομίζω ότι η δικιά μας θέση ήταν ότι πρέπει οι περιφέρειες να συνδιαμορφώσουν τα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης με τα κεντρικά κράτη. Ε, αν καταλαβαίνω καλά από την έκθεση υπονοείται ότι αυτό είναι μια, μια δυσκολία και ότι ε, αυτή η διαδικασία δημιουργεί καθυστερήσεις. Είναι προφανώς χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο για να οργανώσει τη διαβούλευση αλλά νομίζω ότι είναι ο πιο σωστό τρόπος όταν μιλάμε για περιφερειακή ανάπτυξη να συμμετέχουν στα σχέδια και στην, ε, και στη σύμβαση ή συμφωνία εταιρική σχέση οι περιφέρειες. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι αντικίνητρο γιατί έτσι μόνο μπορούμε να έχουμε ισορροπημένα σχέδια περιφερειακή ανάπτυξη. Εγώ δεν το βλέπω καθόλου ως κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται για να έχουμε πετυχημένα δηλαδή αν καταλαβαίνω καλά από την έκθεση υπονοείται ότι είναι καλύτερο τα κράτη μέλη να έχουν μια πιο κεντρική ε, διαμόρφωση των προγραμμάτων τους και όχι πολλά περιφερειακά σχέδια, επιχειρησιακά σχέδια, γιατί αυτό δημιουργεί σύνθετες καταστάσεις και απαιτούνται νέες δομές. Μα όμως νομίζω ότι ο στόχος περιφερειακής ανάπτυξης είναι κυρίως οι περιφέρειες να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός σχεδίου ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά τους, τις προτεραιότητές τους και αυτό να είναι το συνολικό εθνικό σχέδιο, το οποίο προφανώς πρέπει να συνδιαμορφώνεται μεταξύ των περιφερειών και του κεντρικού κράτους και αυτό θα πρέπει να συνυπογράφεται με την ε, Κομισιόν για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Η δυσκολία είναι στο να υπάρχει αυτός ο διάλογος στις χώρες που δεν έχουν ομοσπονδιακή δομή και πράγματι το κεντρικό κράτος να συνομιλεί τα Υπουργεία μεταξύ τους και τα Υπουργεία με τις περιφέρειες. Νομίζω το συντάγαμε και στις προηγούμενες εκθέσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Διάλογος μεταξύ των Υπουργείων, να μην κάνει το κάθε Υπουργείο ένα χωριστό πρόγραμμα, αλλά υπάρχει συνοχή, αλλά και ταυτόχρονα το κεντρικό κράτος να συνομιλεί με τις περιφέρειες και να συνδιαμορφώνει τα σχέδια. Αυτό έχω την εντύπωση ότι δεν έχει προχωρήσει πολύ, εκτός από τις χώρες που έχουν πιο ομοσπονδιακή δομή και είναι καλύτερα προετοιμασμένες για κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον από την, τη δικιά μου χώρα και κάποιες άλλες χώρες που ξέρω δεν έχει γίνει κατανοητό αυτό. Το κάθε Υπουργείο υποβάλλει ένα σχέδιο και σπάνια διαβουλεύεται αναλυτικά με τις περιφέρειες και πολύ περισσότερο και με τους κοινωνικούς φορείς σε κάθε περιφέρεια. Γιατί ε, δεν μιλάμε ενόηση με τον Περιφερειάρχη ή απλώς με ένα Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και με τους κοινωνικούς εταίρους πριν από λίγο συζητάγαμε για την ευφύ εξειδίκευση άρα όλο αυτό είναι πράγματι σύνθετο αλλά πρέπει να αποτυπώνεται στην, σχέση, στην σύμβαση εταιρική ε, σχέσης. Αυτό θα είναι τότε πετυχημένο σχέδιο και θα έχει αποτέλεσμα. Thank you. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θέλει να απαντήσει η Κομισιόν. Παρακαλώ. Καλό απόγευμα. Είμαι από την ε, DG Regio. Ασχολούμαστε πάρα πολύ, είμαστε απολύτως εμπλεγμένοι σε αυτή τη διαπραγμάτευση, γιατί ασχολούμαστε πολύ και με την γεωγραφική κατάτμιση. Όσον αφορά την ίδια την έκθεση, Βεβαίως, θίγει όλα τα απαραίτητα θέματα και εμείς θεωρούμε ότι η έγκαιρη ε, αρχή του, των προγραμμάτων είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις ε, και βεβαίως πρώτα χρειαζόμαστε τους κανονισμούς ε, και μετά την υλοποίηση του χρηματοδοτικού πλαισίου. Και βεβαίως προϋποθέτουμε και την προϋπόθεση συγγνώμη, είναι και η πλήρη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Είμαστε στην ευτυχή θέση να πούμε ότι έτσι όπως φαίνεται η κατάσταση και ήδη και από την, τελευταία χρονιά ε, έχει ξεκινήσει από πλευρά κρατών μελών πολύ εντατικός διάλογος ε, με την ε, Κομισιόν. Δεύτερον, το οποίο αναφέρεται και στην έκθεση, αλλά ίσως όχι τόσο σαφώς, είναι η ποιότητα του προγράμματος ε, και όσον αφορά την σαφήνεια των στόχων και όσον αφορά τη χρηματοδότηση, όσον αφορά τους ρεαλιστικούς στόχους. Αυτά είναι όλα ζητήματα τα οποία τα έχουμε δει σε πολλές περιφέρειες. Εκεί καμιά φορά έχουν δυσκολίες και όλες κάποιες ε, περιφέρειες και θα πρέπει να αποσαφινιστούν μερικά πράγματα ε, περισσότερο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ξεκινήσουμε από την αρχή με καλό ρυθμό έτσι ώστε όχι μόνο έγκαιρα να ξεκινήσουν τα προγράμματα, αλλά να έχουν και καλή ποιότητα τα προγράμματα αυτά, έτσι ώστε να μην είμαστε λαχανιασμένοι προς το τέλος της ε, περίοδου κατά κάποιο τρόπο. Ε, επομένως προγράμματα τα οποία θα είναι σωστά γιατί θα δαπανηθούν και χρήματα σε αυτά τα προγράμματα τα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά την ποιότητα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει στους νέους κανονισμούς ε, η εξάντε, η εκ των προτέρων ερεσιμότητα. εξάντε conditionality. Ε, και προβλέπεται επίσης ε, και πλήρης αξιολόγηση ήδη από την αρχή. Πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ καλά και σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη μέχρι την αρχή του προγράμματος γιατί αυτή η εξάντε conditionality, η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα είναι ακρογωνιαίος λήθος για το πρόγραμμα. Ο λόγος για τον οποίο ορισμένες ε, περιφέρειες ή περιοχές είναι πιο μπροστά και άλλες λίγο πιο πίσω, οι λόγοι λοιπόν Λοιπόν, αναφέρονται σωστά στην ε, έκθεση. Ε, θίγει η έκθεση το ζήτημα ότι η Κομισιόν θα έπρεπε να βοηθήσει περισσότερο τις χώρες μέλη οι οποίες ε, έχουν ακόμα περισσότερες ανάγκες χώρες προγράμματος οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες. Αυτό όμως το κάνουμε ήδη. Δουλεύουμε σε στενή συνεργασία με αυτές τι χώρες μέλη. Έχουμε οργανώσει πάρα πολλά σεμινάρια επί Επίσης έχουμε πολλούς πραγματογνώμονες, εμπειρογνώμονες οι οποίοι δουλεύουν σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Να υπογραμμίσω απλώς ότι εν τέλει ε, το πρόγραμμα είναι του κράτους μέλους. Δηλαδή θα πρέπει να το κατέχουν τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να στεφθεί από επιτυχία. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε, μπορούμε να αναθεωρήσουμε, αλλά, να διορθώσουμε, αλλά η ίδια διατύπωση θα πρέπει να έχει γίνει από τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουμε δει λίγα. Παρ' όλα αυτά διαπιστώνουμε ότι ε, οι ε, συγκεκριμένοι στόχοι τελικά δεν είναι τόσο συγκεκριμένη και τόσο στοχευμένη όσο θα θέλαμε. Ε, θέλουμε ε, στόχους οι οποίοι να είναι βεβαίως ε, φιλόδοξοι, αλλά όχι υπερβολικά φιλόδοξοι, ούτε όμως και πολύ λίγο φιλόδοξοι, δηλαδή να είναι πραγματοποιήσιμοι, υλοποιήσιμοι στόχοι. Ε, και επίσης ε, ε, από τον ίδιο τον κανονισμό απορρέουν και συγκεκριμένες υποχρεώσεις όσον αφορά τη θεματική στόχευση, προγραμματική στόχευση κτλ. Επιτόπου λοιπόν ακόμα πρέπει να γίνει η δουλειά. Όσον αφορά το χρηματοδοτικό εργαλείο, νομίζω ότι όταν θα έχουμε το, τις επιχειρησιακές εταιρικέ σχέσεις, τότε θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στο σημείο αυτό. Εταιρικέ σχέσεις τώρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η σημασία των, ε, αυτών των ε, σχέσεων και είναι πολύ ψηλά στο θεματολογιό μας. Όμως ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν έχουν εγκαθιδρυθεί έτσι καλά αυτά, αυτό το, το εργαλείο και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι εάν ένα πρόγραμμα έχει ε, ξεκινήσει και έχει διατυπωθεί σε στενή συνεργασία με τους εταίρους, ε, τότε ε, θα είναι κτήμα τους και θα είναι σωστή η διατύπωση. Γι' αυτό ακριβώς εμείς προσπαθούμε να επιβλέπουμε και να βοηθούμε τα κράτη-μέλη σε αυτό. Τέλος, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε μέχρι το 2014 για να μην χάσουμε το 2014. Μεγάλη ερώτηση. Ε, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως ε, και ε, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο καθυστέρησε λίγο. Είχαμε γενικώ καθυστερήσεις και παρόλα αυτά όμως είχαμε ανεπίσημο διάλογο. Είδαμε ήδη τα προσχέδια εταιρικών σχέσεων. Εξακολουθούν να φτάνουν και άλλα προσχέδια εταιρικών σχέσεων τα οποία μελετούμε. Νομίζω λοιπόν ότι θα τα καταφέρουμε, Μπορούμε, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από τη δικιά μας πλευρά και θα πρέπει βεβαίως και από την πλευρά των κρατών μελών ε, να παίξουν το παιχνίδι με τον ίδιο αντίστοιχο τρόπο. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω άλλη μια ερώτηση που σχετίζεται με την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, ειδικά τα μεγάλα έργα υποδομών. Γνωρίζω πως ε, διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα αυτή τη στιγμή είναι αντικείμενα επεξεργασία και προετοιμάζονται και συμφωνίες ε, όπως εξηγήσετε, αλλά κάποιες προτεραιότητες είναι προφανές. Ε, προφανείς, με συγχωρείτε. Μεταφορές, είδα τα... και λοιπές υποδομές και οι χώρες προετοιμάζουν αιτήσει για τα μεγάλα έργα κάποιες ε, πιθανώς υποβάλλουν τις αιτήσει ήδη. Η Κομισιόν είναι σε θέση να αξιολογήσει αυτές τις ε, αιτήσει ε, κατά τρόπον ώστε οι χώρες να ξεκινήσουν την εφαρμογή αμέσως, δηλαδή από 1η Πρώτου 2014. Κοιτάξτε, τα μεγάλα έργα προφανώς είναι σαφές στοιχείο και της νέας προγραμματικής ε, περίοδου. Τα μεγάλα έργα... Major, major Είναι μεγάλα, εντάξει, και καλύπτουν κάποιοι. Έχουν κάποιες ε, μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες, αλλά δεν ε, υπάρχουν σε ένα κενό. Πρέπει να προκύπτουν από τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να αναφέρονται στο εθνικό σχέδιο κατά το οποίο είναι ε, μέρος ε, της ε, εξάντε ρεσιμότητας. Οπότε η Κομισιόν πρέπει να μπορεί να εξετάσει ένα μεγάλο αυτό ευθυγραμμίζεται με το στρατηγικό πλαίσιο. Αν υπάρχει το πλαίσιο, ναι, προφανώς τότε τα μεγάλα έργα θα τα εξετάσουμε το συντομότερο δυνατόν. Αλλά πρέπει να δούμε και το πλαίσιο. Σας ευχαριστώ, Βίκτορ Μποστινάρου. Without referring to the χωρίς να θελήσω να αναφερθώ στην εταιρική συμφωνία, γιατί έτσι και αλλιώς είναι κάτι που έχει συζητηθεί επανειλημμένα. Έχω ερωτήσεις για τον τρόπο με τον οποίο είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει κάποια σημαντικά σημεία, σαν παράδειγμα την αποφασιστικότητα και ετοιμότητα των κρατών μελών να ασκήσουν την ολοκληρωμένη αυτή αντίληψη, όπως επίσης It's about και τη χρήση των πολλών ταμείων όταν μιλάμε για τέτοιες επενδύσεις εφιούς τύπου και όταν θέλουμε να, να διαφοροποιήσουμε την επόμενη περίοδο από την παρούσα περίοδο επί τη βάση ε, αυτών που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη λοιπόν σήμερα είναι έτοιμα ή ε, έχουν προετοιμαστεί να ασκήσουν αυτές τις νέου τύπου ε, μορφές δράσης. Δεύτερον, έχουν τη διαχειριστική ικανότητα να το πετύχουν, γιατί χρειάζεται εσωτερικά να διευκρινιστούν ορισμένα θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τους κανόνες επιλεξιμότητας, με την διαχειριστική ικανότητα κτλ. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τομέα αυτό. θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει σήμερα τη διοικητική ικανότητα των χωρών, επαναλαμβάνω. Γιατί αν δεν υπάρξει μια ουσιαστική βελτίωση αυτής της ικανότητας σε χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά τα τόσο περίπλοκα, αν θέλετε, στοιχεία να τεθούν σε εφαρμογές. Σχετικά τώρα με το Connecting Europe. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει κάνει τις νέες προτάσεις. Επί τη βάση όμως των πληροφοριών που έχουμε, ο χρονισμός και οι κανόνες θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν σεβαστοί από τα κράτη-μέλη. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας εξηγήσετε σε τι φάση βρίσκονται οι χώρες αυτές ε, και μπορούν να σεβαστούν τους κανόνες της Επιτροπής για το Connecting Europe και μπορούν να προλάβουν τεράστιες ζημίες γιατί τα κράτη-μέλη θα υποστούν τεράστιες ζημίες αν τελικά δεν μπορέσουν να το σεβαστούν. Και τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να μας δώσει ένα συγκεκριμένο και εφικτό χρονοδιάγραμμα για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν τα προγράμματα Connecting Europe. Κοιτάξτε, ξεπεράσαμε την δυνατότητα να υπάρξουν απαντήσεις σε όλα αυτά. Ε, θα πρέπει να μας απαντήσετε πολύ συνοπτικά. Σχετικά για την χρήση πολλαπλών ταμείων. Αυτό έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στα κράτη-μέλη. Έχουμε προβλέψεις από 17 χώρες να έχουν ένα ή περισσότερα προγράμματα πολυχρηματοδοτούμενα. Σε κάποια από τις χώρες τέτοιου είδους υπάρχουν δηλαδή συνδυασμός του κοινωνικού με άλλα. Ήδη από την περίοδο 2006. Για αυτές τις χώρες σε επίπεδο συντονισμού και διαχείρισης τα πράγματα είναι εύκολα. Έχουμε να κάνουμε με μια επιλογή βέβαια, η χρήση των πολλών ταμείων είναι μια δυνατότητα, δεν είναι μια υποχρέωση. Μπορεί κάποιες χώρες να θεωρήσουν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους προγράμματα, ως εκ τούτου δεν τα προτείνουν. Όπου όμως προτείνουν αντίστοιχα τέτοια προγράμματα και όπου υπάρχει η διαχειριστική, αν θέλετε, δυνότητα των κρατών αυτών να προχωρήσουν, μπορούν ήδη από τις προτάσεις που θα καταβάλουν τον επόμενο χρόνο να αξιολογήσουμε τις δυνατότητες αυτές. Υπάρχουν λοιπόν από τον κανονισμό δυνατότητες και επιλογές για τα κράτη-μέλη να κάνουν προτάσεις για τέτοιου είδους προγράμματα εκεί όπου θα τους είναι ωφέλιμο. Αλλά είπα για 17 χώρες ήδη έχουμε πολλαπλά ταμεία τα οποία ε, στηρίζουν προγράμματα. Για το Connecting Europe θα πρέπει να απαντήσει η Γενική Διεύθυνση MOVE. Πράγματι προκλήθηκε μια καλή συζήτηση, αναφέρεται στον εισηγητή, λέει στον κύριο Βον η Πρόεδρος. Κοιτάξτε, οι εκθέσει ιδίας πρωτοβουλίας δεν έχουν σαν στόχο να δίνουν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που υπάρχουν αλλά νομίζω οι πιο σημαντικές έτυχαν αν θέλετε συζήτησης. Εμείς ε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η κοινωνική, το κοινωνικό ταμείο και τα ταμεία συνοχής και να δούμε πώς θα εξελιχθούν στο μέλλον. Σχετικά με κίνητρα δίδονται στα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θέλω να πω ότι οι μικρότερες συγκεντρωτικές κατά κάποιο τρόπο σε επίπεδο διοίκησης χώρες είναι αυτές οι οποίες έχουν προχωρήσει περισσότερο του είδους τα προγράμματα τα οποία μας ενδιαφέρουν τώρα. Αν όμως τα κράτη-μέλη μπορούν να συνεργαστούν με τις επιχειρήσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τότε τα προγράμματα αυτά θα επηρεάσουν πολύ περισσότερο όπως θα θέλαμε προς την κατεύθυνση που θέλει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι τομεί, ε, ε, αν θέλετε, ενασχόληση με τα θέματα αυτά θα θεωρήσουν ότι τα προγράμματα αυτά μπορούν να τα διαχειριστούν, τους ανήκουν κατά κάποιο τρόπο. Το θέμα δεν είναι, καταλαβαίνω να θέλουμε να ξέρουμε ποιος πάει καλά και ποιος δεν πάει καλά, σαν βαθμολογία πρωταθλήματος ποδοσφαίρου δεν νομίζω ότι είναι εκεί το θέμα. Ήθελα κάποια, αν θέλετε, γενικότερα σχόλια. Κάποια παραδείγματα, σαν παράδειγμα, τα οποία να μας δείχνουν ποιες χώρες πάνε καλά, ποιες δεν πάνε καλά και ποιος είναι ο λόγος που δεν γίνεται αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ποια είναι τα προβλήματα και γι' αυτό τέτοιου είδους εκθέσεις είναι χρήσιμες Έχουμε λίγο χρόνο και ελπίζω με τη συνεισφορά των συναδέλφων μέχρι το τέλος της εβδομάδας να καταστεί η έκθεση αυτή ισχυρότερη. Λοιπόν, προθεσμία είναι η 18η Οκτωβρίου να ζητήσω από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι στο, μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές του επομένου χρόνου, θα θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις του ε, Γενικού Διευθυντή σας για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Και το θέμα επίσης της προετοιμασίας των κρατών μελών να ξεκινήσουν αυτού του νέου είδους προγράμματα. Θα έρθουμε σε επαφή λοιπόν με τους γενικούς διευθυντές. Λοιπόν κλείνουμε το θέμα. Η επόμενη συνάντηση είναι τρεις συνεδριάσεις μισής ημέρας από 27 Νοεμβρίου. Δεν αποκλείεται όμως να έχουμε μια έκτακτη συνάντηση στις αρχές Νοεμβρίου αν τυχόν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και έχουμε κάτι το οποίο θα πρέπει να εγκρίνουμε. Τέλος της συνεδρίασης.